Καλημέρα σε όλους σας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν πρώτα απ' όλα Έχουμε την ε, ημερήσια διάταξη. Έχετε κάποια ερώτηση όσον αφορά την ημερήσια διάταξη, σχόλιο, κανένα από ό,τι βλέπω. Επομένως, εγκρίθηκε η ημερήσια διάταξη. Έχω δύο ανακοινώσεις ε, του Προέδρου. Όχι, δεν έχω τίποτα μάλλον. Ε, και επομένως περνάμε στο τρίτο σημείο, δηλαδή Ευρωπαϊκές Εταιρείες Επιχειρηματικού Κεφαλαίου και Ευρωπαϊκά Ταμεία Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Ε, όπως ε, γνωρίζετε, έχουν υπάρξει κάποιες αντιδράσεις και με, κυρίως όσον αφορά την ε, ε, κατεξουσιοδότηση ε, πράξη. Γι' αυτό είπαμε ότι σήμερα θα κάνουμε μια σχετική ε, συζήτηση. Sorry. Sorry for okay. I am not very... Okay. Είπαμε, είμαστε στο σημείο 3. Sí, Fondo Capital, efectivamente. Este asunto gas... Ναι, είναι αυτό που σας έλεγα. Εταιρείε επιχειρηματικού κεφαλαίου ε, της κυρίας ε, Πιέτη Κάινεν. Όπως γνωρίζετε, ξεκίνησε το 2013 το θέμα αυτό ε, έτσι ώστε να γίνουν με στόχο δηλαδή να γίνουν οι επενδύσεις ε, πιο ε, ελκυστικές. Ε, και προτείνονται λοιπόν μια σειρά αλλαγών έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος αυτός. Θα έχουμε λοιπόν σήμερα μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων στα πλαίσια της Επιτροπής μας και θα δώσω αμέσως το λόγο στην κυρία ε, εισηγητρία, στην κυρία Σύρπα Πιέτη So, Ευχαριστώ πολύ. Όπως ακούσατε, το 2013 τέτοιες ισχύει ο κανονισμός. Ε, μιλάμε για ταμεία τα οποία μπορούν ε, να βοηθήσουν ε, καινοτομίες, μικρές και, μεγα... και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στα πλαίσια της Ευρώπης. Αυτό το χρειαζόμαστε πάρα πολύ όπως γνωρίζετε όλοι γιατί ε, ο υψηλός μακροπρόθεσμος κίνδυνος στις, ε, στα επιχειρηματικά κεφάλαια ε, είναι προβληματικά στην Ευρώπη και επομένως αυτό είναι το ζήτημα. Πώς μπορεί κανείς να καλύψει τις μακροπρόθεσμες επενδυσιακές ανάγκες από τη μία και τις δυνατότητες επένδυσης από την άλλη. Στην παρούσα πρόταση μάλλον η παρούσα πρόταση ε, είναι μέλος του σχεδίου δράσης ε, για την ε, ενιαία αγορά κεφαλαίων και έχει στόχο την διευκόλυνση της, της εξέβρεσης κονδυλίων τα οποία θα μπορούσαν να μπουν στις επενδύσεις η διαβούλευση, ε, η διαβούλευση ε, είχε σαν ε, αποτέλεσμα τις προτάσεις για αλλαγές σε τρία επίπεδα. να αυξηθούν ε, οι εταιρείε οι οποίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν, ε, να γίνει η καταχώρηση του, των ταμείων αυτών πιο εύκολη και, πιο, και κυρίως πιο ε, φτηνή. Οι στόχοι γενικώ είναι σωστοί και μπορούμε να τους προσυπογράψουμε. Θα πρέπει βέβαια να καθοριστούν καλύτερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επίσης ε, θα πρέπει να προχωρήσει και η διαβούλευση με το Κοινοβούλιο γιατί έχουμε την εντύπωση ότι οι δράσεις οι οποίες ε, προτείνονται ε, μπορούν να αυξήσουν πραγματικά τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου στα πλαίσια της ομισματικής Ένωσης. Υπάρχουν και κάποια δευτερεύοντα ζητήματα και υπάρχουν και κάποιες προτάσεις τις οποίες θα μπορούσα να κάνω και εγώ. Πρώτα απ' όλα, το μεγαλύτερο πρόβλημα θα είναι ο τρόπος με τον οποίο θα καταφέρουμε να διαχειριστούμε την έγκριση και την επιτήρηση αυτών των κεφαλαίων στην Ευρώπη τα, τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικές πρακτικές, έχουν διαφορετικούς κανόνες και επομένως είναι πάρα πολύ δύσκολο, εξαιρετικά δύσκολο να δημιουργηθούν πανευρωπαϊκά ε, ε, ταμεία και κεφάλαια ε, εάν θέλουμε πραγματικά να δημιουργήσουμε ε, μια ε, κεφαλιακή ένωση ε, θα πρέπει οπωσδήποτε ε, να εγκριθούν οι διαδικασίες αυτές και σε ευρωπαϊκό επίπεδο μάλιστα. Αυτό είναι ένα σημείο το οποίο ενδεχομένως θα αποτελέσει σημείο σύγκρουσης και με τα κράτη-μέλη και επίσης ε, το ζήτημα είναι ότι η ΕΣΜΑ θα πρέπει να ε, αποτελέσει την αρχή επιτήρησης κατά κάποιο τρόπο και θα πρέπει να καταγράψει τους όρους και τις προϋποθέσεις. Ε, επίσης, η απτή επιτήρηση θα πρέπει να γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε κοινή αρμοδιότητα με τα κράτη-μέλη. Θα δούμε λοιπόν με ποιο τρόπο θα συμφωνήσουν και τα κράτη-μέλη όσον αφορά την επιτήρηση. Έχουμε και κάποια άλλα σημεία τα οποία συζητήθηκαν. Θα πρέπει να πειράξουμε το ε, κατόφλι έτσι ώστε να ε, αναφερθούμε μονάχα σε επιχειρηματίες, σε επαγγελματίες, ε, επενδυτές και επίσης ποιος θα είναι ο τρόπος υπολογισμού του κατοφλίου για τους μη επαγγελματίες το κατόφλι είναι αρκετά ε, υψηλό. Ίσως ε, θα μπορούσαμε να δούμε ένα κατόφλι διαφορετικό από τις 50.000, αλλά θα δούμε. Αυτή είναι η συζήτηση και κάθε συζήτηση, ξέρετε, για τέτοιου είδους ε, επιχειρηματικά κεφάλαια κινδύνου θα πρέπει να ε, συζητιέται ενδελεχώς και με τους ενδιαφερόμενους. Όσον αφορά το μέλλον ε, ερώτημα, θα πρέπει να δημιουργηθεί ε, πραγματικά ένα είδος ταμείου εντός των, του venture capital. Πιστεύουμε ότι το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να προτείνει κάτι σχετικό ε, όσον αφορά την επόμενη αναθεώρηση της Κομισιόν, να το υποβάλει δηλαδή ε, στην Κομισιόν. Από την άλλη πλευρά είναι γεγονός ότι έχουμε αρκετά εργαλεία, το ξέρετε αυτό, στις αγορές που είναι διαθέσιμα ήδη για τους ε, ε, καταναλωτές. Κοιτάξτε, εγώ ε, ε, αν υπάρχει ένα κατόφλι ας πούμε των 10.000 εγώ νομίζω ότι πιο εύκολα ε, θα μπορούσα να επενδύσω έστω και αν υπάρχει κίνδυνος επίσης εάν καταλαβαίνω τον κίνδυνο επίσης θα, μπορούσε, θα μπορούσα να επενδύσω πιο εύκολα σε οτιδήποτε σε καινοτομίες, σε νέα πράγματα σε ηλιακή ενέργεια, σε οτιδήποτε επίσης ε, το, το μακροπρόθεσμο είναι ένα άλλο σημείο. Ε, εάν προετοιμαστεί σωστά ε, και ο κίνδυνος μειώνεται και σίγουρα θα γίνει πιο ελκυστικό για τους επενδυτές. Εγώ καταλαβαίνω βεβαίως ότι είναι αμφιλεγόμενο ε, ε, ζήτημα γιατί υπάρχει αυτό το ζήτημα του κινδύνου ε, και επομένως θα πρέπει να το συζητήσουμε και φυσικά και αυτά τα ιδιωτικά χρήματα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν περισσότερο. Ένα επόμενο σημείο όσον αφορά τους διαχειριστές Πιστεύουμε ότι από τη στιγμή που είναι η ίδια η αγορά θα πρέπει στα διαφορετικά κράτη-μέλη ε, θα πρέπει λέω οι διαχειριστές ε, ε, να έχουν τα ίδια προσόντα και επομένως οι απαιτήσει των κρατών μελών θα πρέπει να είναι παρόμοιες. Επίσης καλύτερη διευκρίνηση όσον αφορά το pre-marketing, το marketing έτσι ώστε τα funds να, έχουν, ε, να μπορούν να κάνουν και τις πρώτες τους διερευνήσεις και σε άλλα ε, κράτη-μέλη πριν ξεκινήσουν ε, να ρίξουν πούμε, τα προϊόντα τους στην αγορά εκεί. Ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τα δημόσια, οι τα δημόσια κονδύλια επίσης μέχρι ένα βαθμό, αλλά θα πρέπει να διευκρινιστεί μέσω του κανονισμού αυτού ότι αυτό το είδος τροφοδότησης ε, των venture capital ε, funds ε, θα, δεν θα θεωρείται κρατική επιδότηση υπάρχουν και κάποια άλλα σημεία τα οποία έχουν συζητηθεί ήδη, αλλά ε, νομίζω ότι καλύτερα είναι να ακούσω τους συναδέλφους, τα σχόλια των συναδέλφων, για να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία... πολύ κύριε Πιετικά. Είναι να κάνουμε ένα γύρο, λοιπόν, να ακούσουμε τους και όλες Πρώτα απ' όλα από τους σοσιαλιστές. Τρία λεπτά γιατί 9.45 πρέπει να ψηφίσουμε και καλό θα ήταν να έχουμε ολοκληρώσει. Η ε, κυρία Μπέρες, ναι, όμω δεν θα έπρεπε να έχουμε πέντε λεπτά ο σκιώδη, τουλάχιστον. Λοιπόν, θα γίνω ο κύριο Κοτσολίνος σήμερα. Και θα ήθελα κυρίω να εστιάσω σε τρία ε, σημεία. Αλλά πριν από αυτό, η έκθεση τη εισηγήτριας, η πρότασή τη συγκεκριμένα, για το κατόφλι για το crowdfunding, δεν ξέρω πώς με RTS θα μπορούσαμε να το ρυθμίσουμε. Να το ξανανοίξουμε, σα είναι μια ερώτηση για την Κομισιόν. Τώρα, τα τρία σημεία στα οποία θα ήθελα να αναφερθεί ο κ. Κοτσολίνο. Και δεν συνηθίζω να μιλώ αγγλικά, αλλά επειδή με, ε, μου έχει δώσει ένα αγγλικό σημείο, μας είμαστε στα αγγλικά, το διαβάζω τα αγγλικά κι εγώ. Εστιάζει λοιπόν σε τρία σημεία. Το πρώτο είναι το άρθρο 10, όπου στην πρόταση της Κομισιόν η ΕΣΜΑ είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό του επίπεδου των ιδίων κεφαλαίων, που πιστεύει ότι αυτό θα πρέπει να θεσπίζεται στον κανονισμό. Και ούτως ή άλλως χρειάζεται και κάποιος χρόνος ε, για να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου. Τα ταμεία θα πρέπει αρχικά να έχουν ένα κεφάλαιο 50.000 ευρώ και το πρόσθετο ε, θα πρέπει να είναι το 1 τέταρτο του παγίου, των παγίων ε, εξόδων. Ε, θα πρέπει επίσης να υπάρχει δυνατότητα άμεσης κινητοποίησης του, των κεφαλαίων αυτών. Είναι χρήσιμη ένα μέθοδος, ενδιαφέρουσα, αλλά βέβαια δεν θα πρέπει αυτό να οδηγήσει σε θέμη το ανταγωνισμό μεταξύ αυτών των ταμείων και το FMD που θα έχουν υψηλότερο κατόφλι. Είναι σημαντικό πάντως να εξασφαλιστεί η επαρκής ρευστότητα. Δεύτερο άρθρο, 16.2, για τα τέλη που λέει πρόταση της Κομισιόν δεν μπορούν να επιβάλλονται από την εποπτική αρχή αυτά τα τέλη αυτής της επιβαρύνσης στην χώρα υποδοχής, αλλά θα πρέπει να υπάρχει εποπτεία σε αυτά τα ταμεία. Και το σχετικό κόστος θα πρέπει να, κόστος θα πρέπει να καλύπτεται. και ότι μπορεί να υπάρξουν και περαιτέρω αποπτικά καθήκοντα, τίθεται το θέμα του ισότιμου πεδίου ανταγωνισμού σε σχέση με χώριους ε, φορείς και γι' αυτό το λόγο πιστεύει ότι καλό είναι πράγματι να αναφέρεται στην πρόταση, μια πρόταση για καθορισμό κάποιων τέτοιων τελών. σε ό,τι αφορά ένα υψηλότερο κόστος. Αυτό θα πρέπει να το δούμε πάρα πολύ προσεκτικά. Έπειτα έχετε το ζήτημα της αναλογικότητας. Σε ό,τι αφορά το διπλό καθεστώς, αυτή είναι μια πρόταση. Ε, σε ό,τι αφορά και τα σήματα 10 eu EU-SEF για να μην είναι μεγάλο το διοικητικό άχθος για τους διαχειριστές. Υπάρχει ένα κατόφλι 13 εκατομμύρια ευρώ. Αναλογικό καθεστώς διαχείρισης. Αν το κεφάλαιο είναι μεταξύ 20 και 500 εκατομμυρίων, ενώ μικρές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου δεν μπορούσαν να χρησιμοποιούν αυτά τα σήματα χωρίς όμως να τους επιβάλλονται σημαντικές επιβαρύνσεις. Αυτό θα δώσει όθηση, θα αποτελέσει ένα κίνητρο για ανάπτυξη αυτής της αγοράς και αύξηση των επενδύσεων. Νομίζω ότι και για το προσπέκτου στην ίδια γραμμή ακολουθήσαμε. Σίγουρα πρέπει να δοθούν κρίματα κίνητρα συγγνώμη, για μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ την κυρία Μπερές. ECR από τον κύριο Καμάλ. Υπάρχει κάποιο άλλο που τον εγκαταστήσει, όχι. Άλντε, κυρία Γκουλάρ. Ευχαριστώ. Εγώ μιλώ στο όνομα τη Κόρα, που είναι στο εξωτερικό. Και ζητά συγγνώμη που δεν μπορεί να είναι σήμερα εδώ. Συμφωνώ ε, με πολλά ποσαλικόρα, αλλά όχι 100%. Το βασικό πρόβλημα τέλος πάντων είναι ο κατακαιρματισμός ε, της ευρωπαϊκής αγοράς. Και ότι υπάρχει και το θέμα των τραπεζικών ε, διαμεσολαβητών εμείς στηρίζουμε την Ένωση Κεφαλαίου Αγορών, οπότε η κόρα λέει ότι καλό θα ήταν με τις νομοθετικές μας πράξεις να επιτρέπουμε περισσότερες διασυνοριακές επενδύσεις και προσφυγή σε νέα μέσα για διαφοροποίηση των πηγών κεφαλαίου. Επιμένει η κόρα ότι είναι σημαντικό και στην φάση των νεοφιών επιχειρήσεων, αλλά και όταν έχουν μεγαλύτερη ισχύ πλέον οι επιχειρήσεις, τα scale scale-ups και εκεί χρειάζονται αρκετά σημαντικό κεφάλαιο όταν βρίσκονται σε φάση ταχείας ανάπτυξης. Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σε αυτή τη φάση συχνά πηγαίνουν στο Silicon Valley για να αναζητήσουν χρηματοδότηση. Αυτό είναι ένα σημαντικό πρώτο στοιχείο λοιπόν, αύξηση κεφαλαίου, ενίσχυση κεφαλαιακή. Ιδίω οι εταιρείε επιχειρηματικού κεφαλαίου και τα ταμεία κοινωνική επιχειρηματικότητα θα μπορούσαν να παρέχουν κίνητρα για όλε τι επιχειρήσει που είναι κάτω από τα 500 εκατομμύρια αυτό το πλαφόν που υπάρχει. Μέχρι στιγμής λίγες είναι οι επιχειρήσεις που έχουν πάρει αυτό το σήμα και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να μα απασχολήσει. Η εκτίμηση αντικτύπου τη Κομισιόν δείχνει επίση ξεκάθαρα ότι σε ό,τι αφορά τα ταμεία που έχουν σήμα ή Ιουβέκα. Είναι πολύ σημαντικό το business cross border. Άρα θα πρέπει η νομοθεσία να επιτρέπει μια πιο ευέλικτη και αναλογική προσέγγιση. Αυτά είναι τα δύο μηνύματα της κόρα. Σας ευχαριστούμε κυρία Γκουλάρ. Παπαδημούλη, το όνομα Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Πιετικάινεν για τη δουλειά που έχει κάνει και για την παρουσίαση που μας έκανε. Να πω ότι θεωρώ χρήσιμες τις ε, συμβολές και τις παρατηρήσεις που άκουσα από την κυρία Γκουλάρ και από την κυρία Μπερές. Ε, ο φάκελος είναι πολύ σημαντικός γιατί εντάσσεται σε μια γενικότερη ανάγκη και συζήτηση που αναπτύσσεται για πολιτικές ανάπτυξης στην Ευρώπη. Ε, και τα δύο ταμεία αυτά είναι μια ευκαιρία η αξιολόγηση των επιδόσεων που υπάρχουν μέχρι τώρα για να δούμε πού υπάρχουν αδυναμίες, πού υπάρχουν προβλήματα, πώς θα πετύχουμε καλύτερες επιδόσεις, πώς θα εντάξουμε τις περιφερειακές οικονομίες, πώς θα επωφεληθούν περισσότερο οι περιοχές, οι περιφέρειες, οι οικονομίες και οι επιχειρήσεις που έχουν περισσότερη ανάγκη ε, από τους, ε, την υλοποίηση των στόχων των δύο ταμείων. Η έκθεση που αξιολογεί τις επιδόσεις μας δίνει ορισμένους ε, αριθμούς απογοητευτικούς. Ε, μέχρι τον Απρίλιο του 2016 ε, τα Ταμείο των Επιχειρηματικών Κεφαλαίων έχουν δημιουργηθεί μόνο 70 ταμεία με στόχο να συγκεντρώσουν σε βάθος δύο εκατοιών, ποσό 4,2 ευρώ και προφανώς αυτές οι επιδόσεις δεν μπορούν να αφήσουν κανέναν ικανοποιημένο αν τους συγκρίνουμε με τους στόχους που έχουν τεθεί. Ε, τα πράγματα με τα ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας είναι ακόμη πιο απογοητευτικά καθώς μέχρι στιγμής υπάρχουν μόνο τέσσερα ταμεία σε όλη την Ευρώπη με συνολικό ενεργητικό 32 εκατομμύρια ευρώ μόνο. Η συζήτηση λοιπόν οφείλει να θέσει επιτάπητος πώς θα μπορέσουν να ενισχυθούν αυτά τα επενδυτικά projects και να αφορούν συγκεκριμένους τομείς και κριτήρια που μέχρι τώρα έχουν μείνει πίσω ε, από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία. Η έκθεση της Κομισιόν για τις επιπτώσεις παρουσιάζει ανάγλυφα ε, ως σημαντικό πρόβλημα το χαμηλό ενεργητικό των ταμείων, τις διασυνοριακές επενδύσεις. Και υπάρχουν και μερικά ερωτήματα με την ευκαιρία αυτής της συζήτησης που πρέπει να θέσουμε. Ποιος έχει πρόσβαση σε αυτά τα ταμεία και τα κεφάλαιά τους. Τι κριτήρια θέτουμε και πάνω από ποιο κεφάλαιο κάποιος, κάποιο όριο έχει πρόσβαση σε αυτά τα ταμεία. Ποιος θα τα διαχειρίζεται θεωρώ ότι τα 500 εκατομμύρια ευρώ ως βάση για το πορτοφόλιο κάποιου επενδυτή ε, είναι αρκετά υψηλό για τα σημερινά δεδομένα, ιδιαίτερα για αρκετές χώρες και περιφέρειες και εκτιμώ ότι ενδεχομένως θα πρέπει να μειωθεί. Επίσης πρέπει να σκεφτούμε πραγματικά είναι στόχος αυτών των δύο ταμείων η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η ενίσχυση της χρηματοδότησής τους, όπως επίσης και πώς επιχειρήσεις με κοινωνικό πρόσημο και προφίλ που εμπεριέχουν μεγαλύτερο ρίσκο μπορούν να στηριχθούν περισσότερο. Συμπερασματικά, είναι σημαντικό να εξετάσουμε γιατί τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Επιχειρηματικού Κεφαλαίου περιορίζονται μόνο σε οκτώ κράτη-μέλη και αν τελικά ο σκοπός για την ενίσχυση των καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των κοινωνικών επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη επιτυγχάνεται, μήπως πάλι μένουν πίσω και έξω από τη δράση αυτών των ταμείων χώρες και περιφέρειες με αυξημένο ρίσκο. Μήπως τελικά οι πόροι αυτών των ταμείων και οι επενδύσεις πηγαίνουν και πάλι στις χώρες και τις περιφέρειες που τις έχουν λιγότερο ανάγκη. Να δούμε με άλλα λόγια την σωστή ποιοτική αξιολόγηση των ταμείων και των προγραμμάτων μέχρι σήμερα που φαίνεται ότι δεν έχει γίνει ουσιαστικά. Έχουμε εξετάσει με σωρευτικά κριτήρια πώς θα γίνεται η παροχή ρευστότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να συνυπολογίσουμε ότι μια επιχείρηση που θεωρείται μικρομεσαία σε μια μεγάλη ισχυρή οικονομία μπορεί να είναι μεγαλύτερη από μια μεγάλη επιχείρηση σε μια μικρή και ασθενέστερη οικονομία. Γι' αυτό τα κριτήρια και τα όρια τόσο του κεφαλαίου όσο και των εργαζομένων πρέπει να επανεξεταστούν με πολύ μεγάλη προσοχή. Και ιδιαίτερα, και κλείνω με αυτό κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να δούμε πώς θα ενισχύσουμε περισσότερο την φωνή των μικρών επιχειρήσεων και των start-ups στην πορεία σχεδιασμού και λήψη των αποφάσεων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Παπαδημούλη. Εξ ονόματος των Πρασίνων, ουδής. Επομένως, περνάμε στην ομάδα διευθυντή, ο κύριος Βάλη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ο συνάδελφος Μαρκοτζάνη είχε ε, υποχρέωση παρουσίας ε, σε άλλη επιτροπή. Παρεμένουν λοιπόν εξ ονόματός του. Σε γενικές γραμμές θεωρούμε ότι αυτά τα εργαλεία είναι οπωσδήποτε πολύ σημαντικά, αλλά όπως και όλο το σύστημα ε, της Ένωσης Κεφαλαιογορών δεν θα, δεν θα λειτουργήσει καλά, γιατί δεν έχουν λυθεί ακόμα γενικής φύσεως οικονομικά προβλήματα. Έχουμε ακόμα αυτήν την κατάσταση ε, νομισματικής ανισορροπίας ε, ε, που προκαλεί ακριβώς ανισορροπίες, προβλήματα τα οποία με τη σειρά τους προκαλούν δυσπιστία στην Ευρώπη και επομένως όλες οι επενδύσεις πηγαίνουν προς χώρες οι οποίες επωφελούνται από αυτήν την έλλειψη ισορροπίας Γερμανία, Ολλανδία κτλ. Ε, ε, επομένως, εμείς πιστεύουμε ότι ε, δεν θα απογειωθούν αυτές οι επενδύσεις. Μην λησμονείτε ότι υπάρχει το θέμα της προσφοράς και της ζήτησης. Δηλαδή, ή θα γίνουν πραγματικές επενδύσεις στην οικοδομία ή δεν πρόκειται να απεμπλακεί η κατάσταση. Ο καλύτερος τρόπος θα ήταν οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης να ξεκινήσουν μαζικά επενδύσεις σε χώρες οι οποίες έχουν πιεστεί. Αλλά ε, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα πρέπει να το αποφασίσει η Γερμανία. Είναι και σε προεκλογική περίοδο τώρα, δεν ελπίζω και πολλά. Ε, όσον αφορά τώρα την ίδια την έκθεση, θα την αναλύσουμε από τεχνική άποψη. Ε, βεβαίως εμείς θα την μελετήσουμε ε, με πολύ θετικό τρόπο. Θα δούμε κυρίως την διαφάνεια και βεβαίως θα θέλουμε εμείς οι επενδύσεις ε, των ταμείων αυτών να γίνουν με διαφάνεια αλλά και προς ε, τις ανάγκες οι οποίες ε, είναι πιο έντονες στην Ευρώπη για νεοφυείς επιχειρήσεις κλπ. Πάντως τα εργαλεία αυτά δεν θα λειτουργήσουν, το ξαναλέω, εάν δεν απεμπλέξουμε την κατάσταση, εάν δεν προχωρήσουμε την κατάσταση όσον αφορά το θέμα της έλλειψης ισορροπίας αφενός και της ενίσχυσης της ζήτησης από την άλλη. Θα πρέπει η Γερμανία να αλλάξει ε, ε, οπτική η οικονομική διαφορετικά η Ευρωζώνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να προχωρήσει. Ευχαριστώ πολύ. Ε, θα, θα δώσω το λόγο στην κυρία Πιτικάινεν ε, σύντομα έτσι ώστε να ολοκληρώσει τη συζήτηση. Thank you. Ευχαριστώ πολύ όλους και όλες. Νομίζω ότι πολλά από αυτά μπορώ να τα συμπεριλάβω και άκουσα ότι εκφράσατε αρκετή υποστήριξη σε ό,τι αφορά ε, το να μπουν 50.000 ευρώ ως κατώτατο όριο ε, που θα το δούμε γιατί νομίζω ότι είναι κάτι θετικό, είναι μια θετική κίνηση. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Πιετικάινεν σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα. 12 Ιανουαρίου θα συζητήσουμε κατάθεση τροπολογιών. Η προθεσμία λίγη 24 Ιανουαρίου, 27 και 28 Ιανουαρίου εξέταση τροπολογιών και προβλέπεται η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας να λάβει χώρα στις 22-23 Μαρτίου και Ολομέλεια Μαΐου. Μαΐου. Υπάρχουν ερωτήσεις? Όχι, ευχαριστώ. Επομένως θα περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο της σημερινής διάταξης. Σας δίνω ένα λεπτό

Dear colleagues, please. Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε. We will start a very important. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες, πολύ σημαντικές όλες. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να κάνουμε έναν έλεγχο. Ε, χρησιμοποιήστε τις ηλεκτρονικές κάρτες σας, βάλτε στο μηχάνημα για να διαλέξουμε τι δουλεύει. Έναρξη του ελέγχου. Because only So, still a lot of people to vote. Ας ψηφίσουν όλοι οι συνάδελφοι που είναι παρόντες, για να γνωρίζουμε. More people to vote. voting card of... Η κάρτα του, του Μάρκος δεν δουλεύει, όχι. Ψηφίσατε αποχή στον έλεγχο, εντάξει. Μάλιστα. Or just some, some Eurobond for... Exactly. Sorry, we, we, got... Συγγνώμη, έχουμε περδευτεί λιγάκι. Τώρα είμαστε ακόμα στον έλεγχο. Ναι, στον έλεγχο, στον έλεγχο. Είμαστε ακόμα. Αλλά αν ψηφίσετε υπέρ, εγώ θα το προσθέσω σε κάποια ψηφοφορία ανάλογα όπως θέλω. Okay, so we close. Μάλιστα, λοιπόν. Κλείνουμε τον έλεγχο, σταματάει η ψηφοφορία. Και ας περάσουμε τώρα στην πρώτη ψηφοφορία επιβεβαίωση για το θέμα των αμοιβαίων κεφαλαίων της χρήματα αγοράς. Πρώτα απ' όλα θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια. Υπενθυμίζοντας τους συναδέλφους ότι η Νατάσα από την Γραμματεία, ιδιαίτερα ικανή συνάδελφος, η οποία μας βοήθησε και ασχολήθηκε με πολλά θέματα ανάμεσα σε αυτόν και για τα ε, αμοιβαία κεφάλαια της χρηματοδορά. είναι η τελευταία της συνεδρίαση και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε και να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε. Θα μας λείψετε. Νίνα, έχετε τον λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ ευχαριστώ και τους συναδέλφους. Μετά από τρία χρόνια καταφέραμε τελικά να καταλήξουμε στη συμφωνία για αυτόν τον κανονισμό για τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματογοράς. Πριν πω οτιδήποτε άλλο θέλω και εγώ να ευχαριστήσω πολλούς. Πρώτα απ' όλα την ομάδα, την διαπραγματευτική, ε, τους σκιώδης, όλους τους συναδέλφους. Ανάμεσα σε αυτούς και εσάς κύριε Πρόεδρε για την συμμετοχή σας. Ήταν μια δύσκολη ε, διαπραγμάτευση, ένα δύσκολο θέμα αλλά με την επιμονή και τη σκληρή δουλειά της γραμματείας, ανάμεσα σε αυτόν και της ε, κυρίας Νατάσα Μάλικ και της Κλόντια, καταφέραμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία που κατά την άποψή μου ισορροπεί τα διάφορες επιδιώξεις, ε, ανταποκρίνεται στις δικές μας ανησυχίες για το συστημικό ρίσκο, αλλά ταυτόχρονα θα καταφέρει να χρηματοδοτήσει την πραγματική οικονομία και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, που είναι και το πιο σημαντικό. Αν έχω το λίγα λεπτά ακόμα στη διάθεσή μου, θα ήθελα να πω ότι καταφέραμε πολλά όσον να αφορά την εισαγωγή του ΙΕΝΕΦ e και μεγαλύτερη διαφοροποίηση στο ρίσκο, καλύτερους κανόνες για την ρευστότητα, ε, Όλα τα θέματα λοιπόν που είχαν απασχολήσει ουσιαστικά το Κοινοβούλιο αντιμετωπίστηκαν και γι' αυτόν τον λόγο πιστεύω ότι θα τύχει υποστήριξη, υποστήριξης των συναδέλφων η πρόταση. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Συλλογαγική Προεδρία για το έργο του στο θέμα αυτό. Thank you, Nina. Indeed, is a very important achievement and you get this. Uh, Ευχαριστούμε, Νίνα. Πράγματι, ήταν μεγάλο κατόρθωμα που καταφέρατε ε, να ολοκληρωθεί αυτή η συζήτηση για ένα θεματικό θέμα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία επί του συμφωνημένου κειμένου με ονομαστική κλίση έναρξη ψηφοφορίας. The vote is closed. Πέρα ψηφοφορίας. 37 υπέρ, 8 κατά, 3 αποχές. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα, πρώτη έκθεση. Έκθεση για την τιτλοποίηση, εισηγητής Πολ Τάγκ. Επίσης σημαντικός φάκελος. Μισό λεπτό λέει ο Πρόεδρος. Amendment 1... Uh, Τροπολογία 109 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβασμός ΕΗ υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική B υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική C υπέρ α, ε, έχουμε, ναι, έχουμε ψηφοφορία κατά τμήματα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική E υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική F FBs υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική I υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική J σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική K υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική L υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική M υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική N υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική O σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός O bis υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, ε, συμβιβαστική P υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική PBS ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική Q υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 467 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική μάλλον τροπολογία 467 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, συμβιβαστική R υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβιβαστική S υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβιβαστική T υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία ε, επί του τροποποιημένου κειμένου με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Vote Πέρας. 44 ψήφοι υπέρ, 4 ε, κατά, μία αποχή. Ψηφίζουμε για το νομοθετικό ψήφισμα, πάλι διονομαστικής κλήσεως, ηλεκτρονικά ε, ψηφίζουμε. Πέρας της ψηφοφορίας. 44 ψήφοι υπέρ, 3 κατά, 2 αποχές. Ψηφοφορία επί της απόφασης εκκίνησης διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο. Πάλι ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. 44 ψήφοι υπέρ, 4 κατά, μία αποχή εγκρίνεται λοιπόν. Συγχαρητήρια κύριε εισηγητά. Now we... Okay, now we move to... Περνάμε, τώρα... Ε, Ε, ε, για την 565 ε, συμβιβαστική υπέρ οι συντονιστές τι είναι υπέρ κατά υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 2 κατά αποχές εγκρίνεται, συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές προφορική τροπολογία. Α, πρώτα το, τη συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία υπέρ. Προφορική υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβιβαστική 7α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία επί του τροποποιημένου κειμένου με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Ε, 40 ψήφοι υπέρ, 9 ψήφοι κατά, καμία αποχή, νομοθετικό ψήφισμα, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ίδιο αποτέλεσμα 49-0. Ε, ψηφίζουμε τώρα για την απόφαση άναξης διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 44 ψήφοι υπέρ, 5 ψήφοι κατά, καμία αποχή. Εγκρίνεται λοιπόν συγχαρητήρια στον εισηγητή κύριο Κάρας. Τώρα τι έχουμε, την πολιτική ανταγωνισμού. Για δώστε μου και τον κατάλογο παρακαλώ. Ευχαριστώ. Okay, ready. Λοιπόν, έχω και τον κατάλογο. Μπορούμε να ξεκινήσουμε στα έτοιμοι. Πέτερ, δεν είναι η σωστή ε, λίστα αυτή που έχω. Μπορείτε να μου φέρετε μια... Okay. Sorry, I found it. Yeah, you have it? Is the last one? I don't know. This is the last one because I had one yesterday. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I'll give you mine. This is the, this is for sure the last one. This is the absolute last one. Okay, so. Λοιπόν. Ετήσια έκθεση σχετικά με την πολιτική ανταγωνισμού. Τσάνισε τη συμβαστική ένα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική B υπέρ, κατά, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολή 69 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 70 υπέρ, κατά, ελέγχουμε την 70, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 71. Υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε την 71 η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Υπήρξε ένα τεχνικό πρόβλημα όμως, οπότε κυρίσω εκ νέου την έναρξη ψηφοφορίας για την 71. Πέρας ψηφοφορίας. Οι 26 ψήφισαν υπέρ, εγκρίνεται. D CDE υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Τροπολογία 92 υπέρ, κατά. Νομίζω ότι εγκρίνεται να ελέγξουμε όμως άρκετη ψηφοφορία γιατί δεν σηκώνεται τα χέρια. Ένα συνάλφος. Δεν έχει ψηφίσει ακόμη. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική F. Ψήφι περ. Κατά απόχέ εγκρίνεται. Συμβιβαστική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 99 ψήφι υπέρ κατά αποχές Νομίζω εγκρίνεται να ελέγξουμε. Θέλετε να ελέγξουμε. Άρχεται ψηφοφορία. Δύο συνάδελφοι να ψηφίσουν που δεν έχουν ψηφίσει ακόμη. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 100. Ψήφι Κατά. Τι ψηφίζουν οι σοσιαλιστές κατά. Υπέρ. Α, πρέπει να ελέγξουν. Ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Προπολογία 101. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική H σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά. Ελέγχουμε το δεύτερο τμήμα, άρχεται ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε το δεύτερο τμήμα. Πηγαίνουμε στην τροπολογία 118. Ψήφι υπέρ. Κατά ποχές, εγκρίνεται. 119 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 120, όχι, καλύπτεται. 121, 121 υπέρ, κατά, ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται συμβαστική I υπέρ Α, υπάρχει τμηματική ψηφοφορία για το social dumping. Δεν το είχα στον κατάλογο. Λοιπόν, πρώτο τμήμα της συμβιβαστικής I. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Να ελέγξουμε το πρώτο τμήμα. Να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ζητήθηκε έλεγχος για το πρώτο τμήμα. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 125 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 126 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 128 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική J. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική J2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική K υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 149 υπέρ, κατά Νομίζω ότι απορρίπτεται να ελέγξουμε καλύτερα. Άρχεται η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Προπλογή 150 υπέρ. 150. Παρακαλώ να σηκώνετε χέρια. Υπέρ. Κατά. Αν την ελέγξουμε. Άρχεται ψηφοφόρη. Πέρασε. Απορρίφθηκε. 151 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε. 151. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 153 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 154 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε. 154 άρχεται ψηφοφορία. Έχετε ψηφίσει όλοι. Συνάδελφοι, παρακαλώ. Λοιπόν, έληξε η ψηφοφορία εγκρίνεται. 155 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική L υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 167 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 171 υπέρ. 171 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε την 171. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 172 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 173 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 174 υπέρ. Κατά να την ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 181. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 179 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 180 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 178 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 182 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική M. Μη. Πρέπει να ψηφίσουμε και το αρχικό κείμενο. Όχι, όχι. Συμβιβαστική M. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ψήφι υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε το πρώτο τμήμα της συμβιβαστικής M. Άρχεται η ψηφοφορία. Vote is closed. Πέρας ψηφοφορία συγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 184 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 186 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 190 υπέρ. Κατά αποχές δεν βλέπω το ΕΛΚ τι κάνει στο 190. Να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε με μία ψήφο διαφορά. 191 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 192 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 193 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 194 υπέρ, κατά ελέγχουμε, άρχεται η ψηφοφορία 191. Εγκρίνεται. ήταν 195, 194 κατά πίπτη, 197 υπέρ, κατά, ελέγχουμε, 197, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε. Μία ψήφος διαφορά. 198 υπέρ. Ελέγχουν. 198. Πέρασε ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε με μία ε, ψήφο διαφορά. Και πάλι. 199 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 200 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε και αυτή 201 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 202 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 203 υπέρ κατά Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά ας ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. 203. Πέρας ψηφοφορίας. εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. 207 υπέρ, κατά, ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία 207. Okay. Vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας. Ο κ. Μακδόναλντ ε, καλά τα κατάφερε. Συμβιβαστική επόμενη, εν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 220 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική ο, ο μικρόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 223 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 225 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 226 υπέρ, κατά, ελέγχουμε. Τη 226 άρχεται ψηφοφορία. Vote is Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 227 υπέρ. Κατά. Το ΕΛΚ δεν βλέπω να ψηφίζει. 227 να ελέγξουμε άρχεται ψηφοφορία. Ήσασταν κατά. Μάλιστα. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 228 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε τη 228 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 229 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ελέγχουμε. Ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Περνάμε στη συμβιβαστική όμικρον 2 με προφορική τροπολογία. Να βλέπω και κανένα χέρι όμως. Λοιπόν, υπάρχουν αντιρρήσεις στην προφορική τροπολογία. Επομένως ψηφίζουμε τη συμβιβαστική χωρίς την προφορική τροπολογία. Ψήφι υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 260 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 249 υπέρ. Κατά αποχές ελέγχουμε τη 249 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. 247 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 251 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 261 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 263 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 265 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 266 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2,77 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε έρχεται ψηφοφορία. Πρέπει να πάμε πίσω. Ξέχασα τη συμβιβαστική π. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα θα ψηφίσουμε τη 277. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 2, 7, 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 283 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 284 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αρχικό κείμενο της παραγράφου 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 285 υπέρ κατά ελέγχουμε τη 285 άρχεται η ψηφοφορία Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 286 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 288 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 292 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 290 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. Ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. 290. Πέρασε ψηφοφορία Απορρίφθηκε. 289 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 291 υπέρ. Κατά ελέγχουμε και 291 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε ψηφοφορίας εγκρίνεται. 2,93 υπέρ. Κατά. Άποχες. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Ας ελέγξουμε όμως. Γιατί δεν σηκώσατε τα χέρια σας. Άρχεται η ψηφοφορία. 2,93. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Μάλιστα. 294 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 297 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 296 υπέρ, κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά ελέγξουμε, άρχεται η ψηφοφορία. Έληξε ψηφοφορία, απορρίφθηκε 2.95 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 2.98 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική Q υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 301 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 302 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 303 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 304 υπέρ κατά. Κατά μάλλον τώρα. Α ελέγξουμε την 304 έναρξη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 305 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 306 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 307 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 308 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 309 υπέρ κατά ας ελέγξουμε την 309 ένα της ψηφορίας για την 309 309 Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 310 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ας ελέγξουμε. Για την 310 λοιπόν, της ψηφοφορίας ηλεκτρονικά. Vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 311 υπέρ κατά. Ε, ας ελέγξουμε ε, έναρξη ψηφοφορίας. Επαναλαμβάνουμε γιατί έγινε ένα λάθος τεχνικό. 311 ηλεκτρονική ψηφοφορία. 311. Ωραία, μπορούμε να κλείσουμε την ψηφοφορία τώρα. Εγκρίνεται. 312. Όχι, έχει καταπέσει. Επομένω, το ίδιο συμβαίνει και για την... Το αρχικό κείμενο 313 υπέρ κατά εποχές. Εγκρίνεται 314 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται 315 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται 316 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Επομένως, καταπίπτουν οι υπόλοιπες. 319 υπέρ κατά αποχές. Ας ελέγξουμε 319. Ψηφίστε παρακαλώ. Vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 320 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 321 υπέρ κατά ας ελέγξουμε 321 έναρξη ψηφοφορίας Vote is closed. ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Επομένως, καταπίπτουν οι υπόλοιπες 327 327 υπέρ, κατά, ας ελέγξουμε, 327. Vote is closed. Εγκρίνεται. 328 υπέρ. 328 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική R, υπές, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 330, υπέρ, κατά, αποχές, ε, απορρίπτεται. 431, υπέρ, κατά. Μάλλον είναι κρίθη, αλλά σε ελέγξουμε για την 331. Πέρας ψηφορίας εγκρίνεται. 332 υπέρ κατά. Ας ελέγξουμε 332, ψηφίστε παρακαλώ. Vote is closed. Πέρα Εγκρίνεται. 333 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε. Ένα της ψηφοφορίας. Πέρασε. Εγκρίνεται. 334 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 335 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 336 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 337 κατά υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 338 συγγνώμη 340 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 343 υπέρ κατά αποχές κατά ε, ας ελέγξουμε καλύτερα 343 Vote is closed. Adopt πέρας ψηφοές ε, συμβαστική S υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα που πάμε Ωραία, συμβαστική τι υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 349 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται 351 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 352 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 353 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 355 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 356 υπέρ κατά Ας ελέγξουμε 356. Ψηφίστε παρακαλώ. Vote is closed. Πέρασε. Απορρίπτεται. 357. Ε, συγγνώμη, 58. Υπέρ κατά αποχέ. Απορρίπτεται. 359. Υπέρ κατά αποχέ. Απορρίπτεται. 361. Υπέρ κατά αποχέ. Απορρίπτεται. 360. Υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. 362 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 363 υπέρ κατά. Ας ελέγξουμε 363 ψηφίστε παρακαλώ. Vote is closed απορρίπτεται. Συμβιβαστική U υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική U2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 365 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 366 υπέρ κατά. Ας ελέγξουμε 366 ψηφίστε παρακαλώ. Vote is Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 368 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε. Έναρξη ψηφοφορίας για να είμαστε σίγουροι. Vote is... Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Με μία ψήφο διαφορά. 369 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 370 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 371 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 372 υπέρ κατά ας ελέγξουμε την 372 ψηφίζουμε στις ψηφοφορίες Εγκρίνεται. 373 υπέρ κατά. Πρέπει να ελέγξουμε. Ψηφίστε παρακαλώ. στις ψηφοφορίες Εγκρίνεται. 374 υπέρ κατά. Ας ελέγξουμε 374. Ψηφίστε παρακαλώ. Εγκρίνεται 375 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε 375. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 377 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε. Λυπάμαι, ορισμένα πολιτικές ομάδες δεν δείχνουν τι ψηφίζουν. 377. Ψηφίστε παρακαλώ. Περιμένουμε. Άμα δεν θέλετε εντάξει. Κλείνουμε την ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 378 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 379 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε. 379. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορία Και κρίνεται. Με μία ψήφο. 380 υπέρ. Ε, κατά. 380 ε, ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορία... Πέρασε Εγκρίνεται. 383 υπέρ. Για τη Φόρμουλα 1. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 384 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 385 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 386 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 387 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 388 υπέρ κατά ας ελέγξουμε ψηφίστε για την 388 παρακαλώ Vote is closed. Εγκρίνεται. 391. 391 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε ψηφοφορία για την 391. Περιμένουμε ακόμα ορισμένου συναδέλφου που δεν έχουν ψηφίσει. 391. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 395 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, απορρίπτεται. 392 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 394 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η επόμενη αφού ψηφίστηκε 392 και εγκρίθηκε η 394 είναι συμβατή, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, μπορούμε να την ψηφίσουμε. Καλά κάναμε. Λοιπόν, εγκρίθηκε η 394, η καταπίπτει 393 και τώρα θα ψηφίσουμε για την 396, σωστά. Υπέρ λοιπόν για την 396 Όμω αφού κατέπεσε η 393, γι' αυτό θέτω στην ψηφοφορία 396. Υπέρ, κατά. Αποχέ, απορρίπτεται. 397, υπέρ, κατά. Αποχέ, απορρίπτεται. 398, υπέρ, κατά. Αποχέ, απορρίπτεται. 399, υπέρ, κατά. Αποχέ, απορρίπτεται. 400, υπέρ, κατά. Αποχέ, απορρίπτεται. 401, υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται, 402 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 303 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 404, συγγνώμη 5 υπέρ κατά Ας ελέγξουμε 405 ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Και εγκρίνεται. 406 υπέρ κατά αποχές απορριπτεται. Συμβιβαστική Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 408 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 410 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 411 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 413 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 415 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 416 υπέρ. Ας ελέγξουμε για την 416, έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 417 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 418 υπέρ Κατά. 418. Ας ελέγξουμε. Ψηφίστε παρακαλώ. Four eighteen. Vote is closed. περα ψηφοφοριας ψηφοφορίας απορρίπτεται. Συμβιβαστική V2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Συγκρίνεται. 422 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 423 υπέρ κατά Ας ελέγξουμε ψηφίστε για την 423 παρακαλώ Vote is closed. Πέρας ψηφορίες. απορρίπτεται 424 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 425 περ. κατά. Ας ελέγξουμε 425 για να είμαστε σίγουροι νόμιζα απορρίπτεται αλλά να είμαστε σίγουροι. Vote is Πέρας Απορρίπτεται με μία ψήφο διαφορά. 426 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 327 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 428 υπέρ κατά. Ας ελέγξουμε ψηφοφορία για την 428. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Πάλι με μία ψηφοδιαφορά. Οι υπόλοιπες καταπίπτουν και πάμε στην 434 υπέρ. 434 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 437 υπέρ. Συγγνώμη. Έχουμε μια προφορική τροπολογία ε, που έχει υποπληθεί επί της 436 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 437 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 438 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 439 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα, να ψηφίσουμε ομού για αυτά που έρχονται από την ΙΝΤΑ. Συμφωνείτε, όχι. Διαφωνούν κάποιοι συνάδελφοι. Δεν μπορούμε να τα ψηφίσουμε όλα μαζί. ΙΝΤΑ 1 υπέρ υπέρ της ε, κατά, εγκρίνθηκε ίντα 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ίντα 3 υπέρ κατά, υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε ίντα 3 ψηφίστε παρακαλώ Vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Μικρή ε, πλειοψηφία. Είναι τα τέσσερα. Καλύπτεται. Είναι τα, είναι τα πέντε υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Είναι τα επτά υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Είναι τα οκτώ υπέρ. Κατά αποχέ. Ας ελέγξουμε. Ψηφίστε παρακαλώ για την ε, τροπολογία ε, οκτώ της ίντα. Vote is closed. Adopted. Inta 9 in favor. υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ίνκο 1. 1 υπέρ κατά αποχές. Ίνκο ε, εγκρίνεται. Ίνκο 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ίνκο ε, 5 υπέρ κατά αποχές. Ε, ελέγχουμε. Ίνκο 5. 5 ηλεκτρονική υπαλήθευση. Πέρας. Εγκρίνεται. Οι υπόλοιπε ε, ΙΜΚΟ θα ψηφιστούν on block μέχρι το 19, μέχρι το 18. Από την 6 μέχρι τη 18 λοιπόν. Όχι, λέει ο πρόεδρος, μέχρι την 11. 6 μέχρι 11. Όχι, μόνο την 7. Κανένας δεν θέλει αμπλόκ. 7. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ΙΜΚΟ 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ΙΜΚΟ 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά αποχές. Νομίζω πως εγκρίνεται. Εγκρίνεται λοιπόν 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, τραν 2, όχι, τραν 1, δεύτερο τμήμα. Τραν 1 υπέρ κατά εγκρίνεται, τραν 2 υπέρ κατά εγκρίνεται. Να ψηφίσουμε μπλοκ μετά τις υπόλοιπες. Τραν. Από την 3 μέχρι πόσο. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 4 υπέρ κατά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 κατά αποχές ε, ηλεκτρονική επαλήθευση τραν 15 ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία είναι σημαντικό, σημαντική ψηφοφορία key vote λέει ο πρόεδρος πέρας και εγκρίνεται τραν 16 υπέρ κατά αποχές υπέρ και το ΕΛΚ ωραία, εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές δεν βλέπω τι κάνουν οι άλλες ομάδες άρχεται η ψηφοφορία επί της τραν 17 Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 19 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 18 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε τώρα να ψηφίσουμε αν μπλοκ τις υπόλοιπες. Μέχρι την 26. Ωραία, 19 μέχρι 26 αν μπλόκ ε, οι υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται, 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 28 υπέρ κατά η ηλεκτρονική επαλήθευση 28 άρχεται η ψηφοφορία. Very good. Is Εγκρίνεται. Άγκρι, αμπλόκ ή όχι, όχι. Α, δεν, είναι, δεν είμαστε όλοι σύμφωνοι επί της άγκρι. Άγκρι ένα, υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση Άγκρι 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Επί της Άγκρι 1. Ψηφίστε! Ψηφίστε λέει ο Πρόεδρος παρακαλώ. Δεν σας βλέπω να ψηφίζετε. Ξανά. Ψηφίστε παρακαλώ για την Άγκρι 1. Λείπουν πολλές ψήφοι. Ωραία, πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Άγκρι 2 υπέρ. Από τη 2 μέχρι την 8 αμπλόκ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 9 υπέρ κατά αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση επί της Άγκρι 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Πέρας. Εγκρίνεται. Τα υπόλοιπα της Άγκρια Block, πολύ ωραία, υπέρκατά αποχές εγκρίνονται. Ε, η ιδεολογική σκέψη 1 υπέρκατα αποχές εγκρίνεται, 2 υπέρκατα αποχές εγκρίνεται. Ε, ήταν η τροπολογία 1, λοιπόν η τροπολογία 2 εγκρίθηκε υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται η 2 τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία τροπολογία 4 θέλετε ηλεκτρονική επαλήθευση πολύ ωραία το ζητήσατε και σας το προσφέρουμε ηλεκτρονική επαλήθευση τροπολογία 4 άρχεται η ψηφοφορία Πέρας και εγκρίνεται η τροπολογία 4, τροπολογία 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 6 υπέρ. Κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Ω, είστε κατά εσείς. Συγγνώμη, έκανα λάθος, λέει ο Πρόεδρος. Να σηκώνετε τα χέρια σας ε, σύμφωνα με αυτά που λέω. Τροπολογία 6, ηλεκτρονική επαλήθευση, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας και εγκρίνεται τροπολογία υπαριθμών 7 υπέρ, υπέρ παρακαλώ υπέρ της 7 κατά αποχές ε, εγκρίνεται σίγουρα αλλά δεν σηκώνετε τα χέρια σας ε, ε, θα πρέπει να κάνω ηλεκτρονική επαλήθευση όπως και τώρα ας πούμε γιατί δεν ήταν σαφές το αποτέλεσμα άρχεται η ψηφοφορία επί της τροπολογίας 7 πέρας της ψηφοφορίας Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Υπέρ. Όχι. Αρχικό κείμενο ε, για τις αιτιολογικές σκέψεις 4 με 6 Τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση από τις τροπολογίες 13 άρχεται η ψηφοφορία. 13, 13, τροπολογία 13. Πέρας της ψηφοφορίας και εγκρίνεται τροπο, αρχικό κείμενο ε, για τις αιτιολογικές 9 10 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 15 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση επί της τροπολογίας υπαριθμών 15 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 21 υπέρ 21 κατά. Ε, άγκρι επί της αιτιολογικής σκέψης 1 υπέρ κατά υπέρ υπέρ αιτιολογικής σκέψης άγκρι. Α, τις τρεις της άγκρια μπλοκ, πολύ ωραία, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία υπαριθμών 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά αποχές δεν βλέπω τι ψηφίζουν οι πράσινοι. Εγκρίνεται. Είναι υπέρ και οι πράσινοι. 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική W υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβιβαστική Y υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, τροπολογία 37 υπέρ κατά ε, έλεγχος επί της τροπολογίας 38 πέρας εγκρίνεται συμβιβαστική Z υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 45 δεν την ψηφίζουμε, είναι ταυτόσιμη. Τροπολογία 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 48 υπέρ κατά αποχές η Άλντε είναι υπέρ ή κατά, εν πάση περιπτώσει, ηλεκτρονική επαλήθευση επί της τροπολογίας 48. Παρακαλώ. Ψηφίστε. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται Αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 51 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση επί της 51. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. απορρίπτεται λόγω ισοψηφίας 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 53 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση επί 53 άρχεται η ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται Άγκρι, ομπλοκ, από κοινού όλες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Τελική ψηφοφορία επί του κειμένου όπως έχει τροποποιηθεί, ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται. Πέρας της ψηφοφορίας, 33 ψήφοι υπέρ, 6 ψήφοι κατά, 5 αποχέσεις Συγχαρητήρια κύριε Ισηγητά. Please, take the floor. Θέλετε το λόγο κύριε Σιγητάνε. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομα. Ε, πιστεύω ότι αυτό ήταν ένα από τα πιο σημαντικά και δύσκολα θέματα αυτής της χρονιάς και είμαι πραγματικά ε, ευγνώμων προς όλους τους συναδέλφους. Όλοι οι συνάδελφοι συνέβαλαν στην έκθεση. Υπάρχουν τρία κεντρικά θέματα, σημεία τα οποία καλύπτονται από αυτήν την έκθεση. Πρώτα απ' όλα κάναμε σημαντικά βήματα έτσι ώστε ε, να αναγνωρίσουμε ότι ότι η δικαιοσύνη είναι σημαντικό τμήμα των κανόνων της πολιτικής ανταγωνισμού. Δεύτερον, όσον αφορά την ψηφιακή αγορά, κάναμε βήματα προς τα εμπρός. Και τρίτο και ίσως και ακόμα πιο σημαντικό, είναι ότι αναφερθήκαμε στην σωστή πρόοδο της συνεταιριστικής και συνεργατικής οικονομίας. Το θέμα της αηφορίας και των κοινωνικών αξιών είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης είμαι ιδιαίτερος ευγνώμων προς τις, τις επιτροπές του Κοινοβουλίου μας οι οποίες συνέβαλαν τα μάλα και βεβαίως ε, Μάσιμο Κολόμπο, ο Μάσιμο Κολόμπο από την ε, ε, Γραμματεία καθώς επίσης και ο ειδικό μου εμπειρογνώμονας με βοήθησαν πάρα πολύ. Τους ευχαριστώ όλους. Okay. Take the plane at six, so I'm a bit. Morning. you just couldn't So, dear colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι, ήταν μακρά αυτή η ψηφοφορία, αλλά παρακαλώ να ξανακαθίσετε. Dear colleagues, a great pleasure Αγαπητοί συνάδελφοι, με πολύ μεγάλη χαρά καλωσορίζω τον Σλοβακό Υπουργό Οικονομικών και Προεδρεύοντα του ΕΚΟΦΗΝ, τον Πέτερ Κάζιμιρ. Σα ευχαριστούμε πολύ που δεχθήκατε την πρόσκλησή μα να έλθετε εδώ και να μα παρουσιάσετε τις απόψεις σε σχέση με τα επιτεύγματα τη Σλοβακικής Προεδρία στον τομέα που αποτελεί παιδερμοδιότητα τη Επιτροπή ΕΚΟΝ. Ήταν μια πολύ επιτυχη Προεδρία. Παρακαλώ. Ησυχία. Με Πολύ χαρά επίσης ανακοινώνω ότι χθες έγινε ένα επίσης πολύ σημαντικό βήμα προς τα εμπρός με την πολιτική συμφωνία που επετεύχθη στον τριμερή διάλογο για τον κανονισμό περί του προσπέκτους. Πολύ σημαντικό βήμα για τη δημιουργία της Ένωσης Κεφαλαίου. Σήμερα ψήσαμε την τυλοποίηση, άρα προχωράμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσάς και την Προεδρία σας. για την εξαιρετική συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Α, να σας πω ότι ψηφίσαμε και ένα κάτι άλλο πολύ σημαντικό για τις χρηματαγορές, τα αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγορών. Και αυτό είναι σημαντικό. Προχωρούμε λοιπόν με την νομοθεσία μας και μπορεί να ξέρετε επίσης ότι και το Συμβούλιο την Τρίτη κατέληξε σε συμφωνία για το FC2. Πολύ σημαντικό και αυτό. Και βέβαια τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα, ελπίζοντας να καταλήξουμε σε θετικό αποτέλεσμα. Σήμερα λοιπόν έχουμε και τον ε, οικονομικό διάλογο στο πλαίσιο της Οικονομικής Νομισματικής Ένωσης. Οπότε για μια ακόμη φορά θέλω να σας ευχαριστήσω, να σας ευχαριστήσω και προσωπικά γιατί είχατε πολύ καλή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο εξάμεινο αυτό και σας δίνω αμέσως στο λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας δώσω και εγώ συγχαρητήρια γιατί ψηφίσατε το, το ε, πολύ σημαντικό αυτό ε, τη σημαντική έκθεση για την τιτλοποίηση, ένα σημαντικό με προς τα εμπρός. Μετά τη χθεσινή συμφωνία για το προσπέκτους και τη σημερινή ψηφοφορία σας για την ε, τιτλοποίηση, νομίζω ότι έχουμε κάνει για την ε, Ένωση κεφαλαιαγορών ε, σημαντικά βήματα. Πολύ σημαντικές αυτές οι δύο ημέρες λοιπόν. Χαίρομαι που ξαναβρισκόμαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή ΕΚΟΝ, ουσιαστικά για να κλείσω τον κύκλο της Σλοβακικής ε, Προεδρίας. Είναι η τελευταία μου φορά ως Προέδρου του ΕΚΟΦΗΝ. Θα ήθελα να σας αναφέρω τα θέματα που είχαμε στο θεματολόγιο ε, του ΕΚΟΦΗΝ, τα οικονομικά και χρηματοπιστωτικά θέματα. Το δεύτερο ήμιση του έτους ε, πιστεύω ότι σωστά μπορούμε να πούμε ότι είχε κάποιες πολύ σημαντικές ε, στιγμές ε, όπου ε, θα μετασχηματίσουν, θα μεταμορφώσουν την Ένωση και είμαι διπλωματικός στις εκφράσεις μου. Η Ένωση ευτυχώς μέχρι στιγμής είναι ανθεκτική αλλά μακροπρόθεσμα δεν ξέρω κατά πόσο έτσι επιτυγχάνεται η ανάπτυξη και η σταθερότητα. Ε, υπάρχει ακόμη αβεβαιότητα σε ό,τι αφορά τις οικονομικές προοπτικές, το Brexit, έχουμε τις υπερεκλογές του χρόνου, πρόσφατες εξέλιξεις στην Ιταλία, αλλαγή σκητάλης ε, στην Αμερική. Θα χρειαστεί χρόνος για να δούμε Ποιο ήταν ο αντίκτυπο όλων αυτών στην Ευρώπη. Στη διάρκεια τη Σλοβακική Προεδρία προσπαθήσαμε να βαδίσουμε με σταθερά ασφαλή βήματα. Είχαμε πολλά θέματα να συζητήσουμε. Θέλαμε όμω να σπάσουμε για κάποια στερεότυπα στο Συμβούλιο, κάποια ταμπού και να έχουμε μια δομημένη συζήτηση για το μέλλον τη Ευρώπη και ιδίω ό,τι αφορά την εμβάθυνση τη ΟΝΕ. Θέλουμε μεταρρυθμίσεις ε, διαρθρωτικές ε, και πρέπει να τα ολοκληρώσουμε σε επίπεδο ΕΚΟΦΗΝ. Εμείς εστιάσαμε κυρίως ε, στο πολιτικό μείγμα επενδύσεις, μεταρρύθμιση διαρθρωτικών ταμείων και υγιείς ευρωστές χρηματοοικονομικές πολιτικές. Ίσως να διαφοροποιούνται σε σχέση με το πού θα δοθεί περισσότερη έμφαση, γιατί ουσιαστικά η ουσία παραμένει ίδια. Ξέρετε τώρα ότι ένα από τα σημαντικότερα, βασικότερα θέματα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε ήταν διαδικασίες περιβολικού ε, λύματος για Ισπανία-Πορτογαλία. Η Κομισιόν έκανε το καλοκαίρι μια εκτίμηση και είπε ότι αυτές οι δύο χώρες δεν είχαν εφαρμόσει ε, δεν είχαν εφαρμόσει ικανοποιητικά τις προτάσεις. Και έπρεπε ότι είπε η Κομισιόν να επιληφθεί και κάποια πρόστιμα στις δύο χώρες. Ε, το Συμβούλιο δεν φαίνονταν να θέλει να διαφοροποιηθεί σε ό,τι αφορά αυτή την προσέγγιση. Εσείς είχατε διαρθρωμένο διάλογο με την Κομισιόν. και με τους Υπουργούς Οικονομικών των δύο χωρών Ισπανίας Πορτογαλίας είχατε επαφέ. Δεν ήταν πάντοτε και σε εμά σαφές το Συμβούλιο περί πρόκειται. Υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις. Πάντως ε, με την ενεργοποίηση αυτής της διαδικασίας ε, οι δύο χώρες κινητοποιήθηκαν και αυτές έλαβαν μέτρα και αυτό ήταν και το αποτέλεσμα τελικά της όλης διαδικασίας. Άρα είχαμε happy end στο τέλος. Και αυτό είναι το καλό και το σημαντικό. Σε ό,τι αφορά τώρα την δημοσιονομική σταθεροποίηση. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε σταθερά δημόσια οικονομικά και να είμαστε αξιόπιστοι. Άρα είναι σημαντική η σταθεροποίηση και βέβαια η δημοσιονομική πολιτική θα πρέπει να έχει στόχο και τη μακροοικονομική σταθεροποίηση. Στο ECOFIN, στο Eurogroup συζητούνται οι προτάσει της Κομισιόν για τη δημοσιονομική ικανότητα τη Ευρωζώνης και όλα αυτά δείχνουν πόσο πολύπλοκο είναι αυτό το ζήτημα. Δείχνει επίση όλη αυτή η συζήτηση ότι οι δημοσιονομικοί κανόνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχαν γνώμονα ε, τη μακροοικονομική σταθερότητα. Και πραγματικά αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο είπε η Σλοβακική Προεδρία ότι αυτή αποτελεί μια από τι βασικέ μα πολιτικέ προτεραιότητε. Δηλαδή να εμβαθύνουμε την ΟΝΕ, να ε, συζητήσουμε όμω ε, το δημοσιονομικό πυλώνα σε επίπεδο υπουργικό. Στη Βρατισλάβα λοιπόν το Σεπτέμβριο έγινε αυτή η συνάντηση και η συζήτηση εστίασε στην δημοσιονομική ικανότητα της Ευρωζώνης πώς θα προστατευτούμε από μακροοικονομικούς κραδασμούς ήταν ένα άλλο θέμα και πραγματικά σπάσαμε ταμπού ε, που για πολλούς ή κάποιους τέλος πάντων ε, στο Συμβούλιο ήταν θέματα που δεν συζητούνταν. Οι Υπουργοί Οικονομικών θα έλεγα ήταν πολύ επικοδομητικοί στην προσέγγισή τους. Βάλαμε επίσης το θέμα στην μέση για διάταξη του ΕΚΟΦΗ του Δεκεμβρίου για αυτή τη βδομάδα γιατί θέλαμε η πρωτοβουλία αυτή να μείνει ζωντανή και να δούμε και τι θα, ποια θα είναι η συνέχεια που θα δώσει η Κομισιόν στην έκθεση των πέντε Προέδρων. Είχαμε τη Λευκή Βίβλο για το μέλλον της Ευρώπης ε, το Μάρτιο, περιμένουμε να δημοσιοποιηθεί και βέβαια θέλουμε να δούμε και τι θα γίνει με τη μελλοντική αρχιτεκτονική της ΟΝΕ. Τον Ιούλιο είχαμε μια ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων για το θέμα αυτό με ευρωβουλευτές και τους υπουργούς οικονομικών. Θέλω να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο διότι διαφώτισε και αυτό με τη δική του συμβολή αυτό το πολύ σημαντικό θέμα και ελπίζω να συνεχίζετε τις δραστηριότητές σας και τις εργασίες σας επ' αυτού. Σίγουρα υπάρχουν διαφορές, υπάρχουν αποκλήσεις, πάντως υπάρχει σε συμβούλιο, στο Συμβούλιο συμφωνία ότι η ΟΝΕ ναι ακόμη δεν είναι παρκώς ανθεκτική. Άρα πρέπει να γίνουν περισσότερα πράγματα. Και ελπίζω ότι στο τέλος του 2017 με τις ε, υπερεκλογές, το, τις σούπερ εκλογές που έχουμε, θα έχουμε επιτύχει σημαντική πρόοδο και με τη βοήθεια της Κομισιόν. Έρχομαι στις επενδύσεις. Επίσης πολύ σημαντικό θέμα για εμάς. Και νομίζω ότι η πρόοδος ε, στον τομέα αυτό είναι αξιοσημείωτη. Το Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ ε, υιοθέτησε τη γενική προσέγγιση για το ΕΦΣΙ 2 και στις 6 Δεκεμβρίου, την Τρίτη συγκεκριμένα, εγκρίναμε αυτή τη γενική προσέγγιση του Συμβουλίου στο ΕΚΟΦΗΝ. Άρα, και ε, επιμικίναμε τον κύκλο ζωής του Ταμείου, αλλά βελτιώσαμε ταυτόχρονα και τις ποιοτικές του πτυχές. Προσθετικότητα, γεωγραφική τομεακή κάλυψη, εστίαση στη δράση για το κλίμα Επίσης ο κόμβος για την παροχή συμβουλών, ευρωπαϊκό κόμβο συμβουλών, πολύ σημαντικό αυτό το hub. Άρα μεγαλύτερος κύκλος ζωής για το ΕΦΣΥ και βελτιωμένη επενδυτική στόχη. Πιστεύω ότι αυτό θα δώσει μεγαλύτερο δυναμικό, θα αναζωογονήσει το Ταμείο. Είμαι πεπισμένος ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να διευκολύνει μια γρήγορη διεκπαιρέωση του ζητήματος και ελπίζω οι διαπραγματεύσεις σε επίπεδο τριμερούς διαλόγου να προχωρήσουν τάχιστα και στο πλαίσιο της επερχόμενης Προεδρίας. Για τις επενδύσεις θα ήθελα να προσθέσω και κάτι ακόμη. Είναι εξαιρετικό το επενδυτικό πρόγραμμα, το είπα τον Ιούλιο στην Επιτροπή σας άλλωστε, έχουμε και την μετανάστευση ως μεγάλη προτεραιότητα και αυτό πριν καν ξεκινήσει η Προεδρία μας. Χαίρομαι λοιπόν που ολοκληρώθηκαν θετικά και για τους τρεις φακέλους του πακέτου η διαπραγματεύση σε επίπεδο Συμβουλίου. Και για το Ταμείο και για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης. Και τώρα να προχωρήσω στα τραπεζικά ζητήματα, στην Τραπεζική Ένωση. Πώς έχει η κατάσταση λοιπόν είναι σημαντικό να ολοκληρωθεί η Τραπεζική Ένωση. Και για τις προηγούμενες και για τις μελλοντικέ προεδρίες. Εμείς ε, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε πάνω στον οδικό χάρτη που ενέκρινε το Συμβούλιο φέτος τον Ιούνιο. Σίγουρα η συζήτηση δεν είναι εύκολη. Έπρεπε να βρούμε σωστή ισορροπία μεταξύ όλων των πτυχών σε ό,τι αφορά την εγγύηση των καταθέσεων, εμείς δίδαμε σε τεχνικό επίπεδο όλες τις προτάσεις, ε, σε ό,τι αφορά τις κρατικέ χρηματοδοτήσεις, ε, προσχώρηση, αποχώρηση, από έτσι και τα λοιπά. Και έχουμε και την πρόταση της Κομισιόν ε, της προηγούμενης εβδομάδας, θα τα ακούσουμε και την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Θα συνεχιστεί λοιπόν η τεχνική συζήτηση και αυτό μάλιστα ήδη από αύριο, για να μην χάνουμε χρόνο. Επίσης υπάρχουν ε, πλέον οι προϋποθέσεις για να συζητήσουμε τα περί του ενιαίου μηχανισμού εκαθάρισης και το backstop ε, mechanism. Δώσαμε εντολή να ξεκινήσει τις εργασίες του ΙΦΕΣΗ. Ένος κεφαλαίου This, uh, Κάποιοι έχουν αμφιβολίες, ιδίως ό,τι αφορά τους Βρετανούς που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όμως, μην πατάστε. Εμείς θέλουμε το συντομότερο δυνατό να προχωρήσουμε. Ε, όχι όμως κατά τρόπο που να γυρίσει μπούμεραγκ. Δεν θα πρέπει να κάνουμε επιβιασμένε κινήσει ό,τι αφορά την Ένωση Κεφαλαίου Αγορών. Πάντως πρόκειται για κάτι πολύ θετικό που θα δώσει νέα πνοή σε πολλούς επιχειρηματίες. Χθε είχαμε μια συμφωνία για τον κανονισμό ε, προσπέκτου, ε, χθε το βράδυ, που είναι ο πρώτος σταθμό ε, για την Ένωση Κεφαλαίου Αγορών και ένα σημαντικό βήμα προς την ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαίου Επίσης πήραμε το Δεκέμβριο εντολή για το πακέτο για την τίτλοποίηση, τα γνωρίζετε όλα αυτά βέβαια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε σήμερα, όπως μας είπατε, το θέμα, ψήφισε για την τιτλοποίηση. Σας ευχαριστώ πολύ για ένα χριστουγεννιάτικο δώρο που κάνατε και σε εμά και στην Ένωση Κεφαλαίου Τέλος. Σε επίπεδο ομάδων εργασίας έχουμε ήδη συμφωνήσει για τα ευρωπαϊκά ταμεία, για τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου και τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας και τα project θα εγκριθούν επισήμως σε επίπεδο κορεπέρ την επόμενη εβδομάδα. Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Τον προηγούμενο μήνα και μετά από εντατικές διαπραγματεύσεις, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία για ένα σχέδιο κανονισμού για τη δημιουργία ενός ρυθμιστικού πλαισίου για τα κεφάλαια χρηματαγορών. Πολύ σημαντικό θέμα. Μετά την έγκριση, την επίσημη έγκριση χθε σε επίπεδο Συμβουλίου στο Κορεπέρ, έχει γίνει ένα σημαντικό βήμα και σήμερα η ΕΚΟΝ έκανε ένα ακόμη σημαντικό βήμα, ψηφίζοντας σχετική έκθεση. Οι συνομοθέτες λοιπόν έχουν συνεισφέρει σημαντικά στην αύξηση της ε, χρηματοοικονομική και σας ευχαριστούμε. Το Συμβούλιο το Νοέμβριο συμφώνησε τη διαπραγματευτική εντολή σε σχέση με την ενημέρωση των καταναλωτών για τον ψηφιακό κανονισμό και η Μαλτέζικη Προεδρία θα προσπαθήσει να καταλήξει πολιτική συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύντομα, σε αρχέ του επόμενου έτου. Η δική μα Προεδρία δουλεύει σκληρά για να υπάρξει συμφωνία στη διαπραγματευτική εντολή του Συμβούλου για την αναθεώρηση της τέταρτης οδηγίας για το ξέπλυμα χρήματος. Έχουμε χρόνο πριν ολοκληρωθεί η δική μας Προεδρία και γνωρίζω ότι η καταπολέμηση του ξεπλήματος χρήματος και της ε, χρηματοδότησης της τρομοκρατίας είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα και για το Κοινοβούλιο και για το Συμβούλιο. Εγώ είμαι αισιόδοξο. Ελπίζω ότι και τα δύο θεσμικά όργανα θα ε, καταλήξουν σε πολιτική συμφωνία του χρόνου, το συντομότερο δυνατό. Και το κερασάκι στην τούρτα, τα φορολογικά ζητήματα, Φοροαπάτη απάτη. Ήταν προτεραιότητα για την Προεδρία μας και για το ΕΚΟΦΗΝ. Έχουμε πετύχει πράγματα που αντικατοπτρίζουν αυτό. Παραδείγματος χάρη, άμεση φορολογία. Είχαμε σημαντικά αποτελέσματα για τα κριτήρια και τις διαδικασίες για τον κατάλογο των μη συνεργαζόμενων χωρών. Μαύρο κατάλογο το λένε τα μέσα ενημέρωσης. Έχουμε την ομάδα κώδικα συμπεριφοράς για επιχειρήσεις και φορολογία θα μελετήσει όλες αυτές τις χώρες το 2014. Ό,τι αφορά τώρα το έγγραφο του Παναμά, προχωρήσαμε στο ΕΚΟΦΗΝ τροποποιώντας την οδηγία περιδικητικής συνεργασίας για φορολογικά ζητήματα. Οπότε οι φορολογικές αρχές πλέον μπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν την ομοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και σε ό,τι αφορά τα Panama Leaks. Φορολογική διαφάνεια λοιπόν, ανάγκη να καταπολεμηθεί η συγκάλυψη κονδυλίων, κεφαλαίων και η πιο καλή συνεργασία με τις φορολογικές αρχές. Αυτή είναι η στόχη μας και πιστεύω ότι με τον τρόπο αυτό θα καταπολεμήσουμε την ε, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, τη φοροαπάτη, τη φοροδιαφυγή κτλ. Επίσης, πρόσφατα Μελετήσαμε την πρόταση της Κομισιόν για ένα ισότιμο πεδίο φορολογικού ανταγωνισμού. Υπάρχουν τέσσερις φορολογικές προτάσεις. Έχουμε το θέμα επίλυσης φορολογικών διαφορών, την ενιαία, έδρα, ε, την ενιαία βάση, φορολογική βάση για τις εταιρείες και το Δεκέμβριο, την Τρίτη συγκεκριμένα, το ΕΚΟΦΗΝ σημείωσε μεγάλη πρόοδο σε ό,τι αφορά τη γενική αντιμετώπιση κάποιων υβριδικών αναναντιστοιχειών. <coughs> Ήταν ένα θέμα που το πήραμε την προηγούμενη Προεδρία Νομίζω ότι το 95% της οδηγίας το έχουμε πλέον σταθεροποιήσει και άρα θα μπορέσει να εγκριθεί του χρόνου. Φυσικά θέλουμε και την άποψη του ε, Κοινοβουλίου. Έμεση φορολογία. Έχουμε συμπεράσματα για βελτιώσεις στους κανόνες ΦΠΑ για τις ε, συναλλαγές όπου καλύπτονται πτυχές που αφορούν τη βελτίωση των ε, σημερινών κανόνων ε, για το ε, ΦΠΑ. Το ΕΚΟΦΗΝ επίσης σημείωσε την πρόοδο των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής και Νορβηγίας, κάτι καινούριο. Ομόφωνα εγκρίθηκαν από όλα τα κράτη-μέλη τα κείμενα της Σλοβακικής Προεδρίας ως πιθανή των διαπραγματεύσεων. Η Σλοβακή Προεδρία επίση κατέληξε σε συμφωνία για τα συμπεράσματα του Συμβουλίου στο θέμα των ειδικών φόρων κατανάλωση για το αλκοόλ και τα αλκοολούχα ποτά και θα έχουμε την πρόταση του χρόνου για αυτό το θέμα. Και τέλος, φορολογία πάντα. Είχαμε ανταλλαγή απόψεων στο Συμβούλιο για το κατά πόσον η απάτη ε, με το ΦΠΑ θα πρέπει να ενταχθεί στο πεδίο του λεγόμενου ΠΙΦ, τη οδηγία ΠΙΦ. Είναι θέμα του Συμβουλίου Δικαιοσύνη Εσωτερικών Υποθέσεων βέβαια. Χαίρομαι γιατί μετά από πολύ καιρό αναστήθηκε αυτό το θέμα και ξανασυζητείται. Τέλος, δύο λόγια για τον προπολογισμό, για του χρόνου και με αυτό θα ολοκληρώσω. Είναι ένα θέμα που δεν εμπίπτει βέβαια εντελώ στην δική σα αρμοδιότητα, όμως θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ των θεσμικών οργάνων στην διαδικασία συνδιαλλαγής σε ό,τι αφορά το προπολογισμό του 2017 και σας ευχαριστούμε. Είμαι πεπισμένο ότι ο προπολογισμό ε, είναι εύρωστος, δείχνει αλληλεγγύη και νομίζω θα διασκεδάσει τις ανησυχίες των πολιτών, κυρίως για τη μετανάστευση, εσωτερική εξωτερική ασφάλεια, ανάπτυξη και απασχόληση. Κάτι πολύ σημαντικό και για το Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. Uh, for... Εμείς σας ευχαριστούμε για αυτή την ενδιαφέρουσα παρουσίαση που καταδεικνύει πόσο πολλά έγιναν κατά τη διάρκεια της Σλοβακικής, Σλοβακικής Προεδρίας. είχατε σημαντικές επιτυχίες και θα δώσω το λόγο στον κύριο Μπούλτς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη Υπουργή Οικονομικών της Σλοβακίας. Πρώτα απ' όλα εξ ονόματος ομάδος του ΕΛΚ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία που είχατε με μας ε, ως Προεδρεύων του Συμβουλίου Κοφίν. Κάνατε πολύ καλή δουλειά και εσείς και οι συνάδελφοί σας ε, και συνεργάτες σας κάνατε κάποιες εκτιμήσεις για την κατάσταση της Τραπεζικής Ένωσης και θα ήθελα να επανέλθω σε αυτό για να σας ζητήσω να μου πείτε κάτι πιο συγκεκριμένο σε ό,τι αφορά την ιδέα ενός ε, συστήματος εκεί των ε, καταθέσεων, το έντις. Κατά την άποψή μου, δεν έχει γίνει μια γενική μελέτη ε, σκοπιμότητας και αντικτύπου. Μέχρι στιγμής ε, η Κομισιόν έχει κάνει μόνο μία τεχνική ανάλυση. Η πρόταση για το έντις ε, επίσης δεν ε, συνδέει τις προτάσεις αυτές με τις προτάσεις μείωση των κινδύνων. Το αναφέρατε για το τραπεζικό τομέα. Υπάρχουν κάποια βήματα για μείωση των κινδύνων αλλά δεν, έχει δείξει, ε, δεν έχουν δείξει συναδελφοί σας οι να επαρκή φιλοδοξία στον τομέα αυτό. Στο μέλλον πρέπει να γίνουν σημαντικά βήματα, γρήγορα βήματα στο έντις. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι κάτι απόλυτα εφικτό. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε κύριε Κάζιμιρ με την απόψη μου ότι η πρόταση έντις ε, υπό τη μορφή που την έχει προτείνει η Κομισιόν ε, μάλλον έχει αποτύχει ή τέλος πάντων θα πρέπει να τροποποιηθεί σημαντικά. Συμφωνείτε ότι αυτό πρέπει να γίνει από πλευρά Κομισιόν, μια ριζική αλλαγή αυτού του κανονισμού. Let me answer in my native language. Θα μιλήσω στη μητρική μου. Σας ευχαριστώ. Ξεκινώ από τον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Όπω θα θυμάστε, ε, στη συνάντησή μα τον Ιούλιο είχαμε μιλήσει για το ΕΔΙΣ και είχα υπάρξει πολύ προσεκτικό στη διατύπωσή μου γιατί πράγματι στο Συμβούλιο έχει γίνει μια έντονη συζήτηση όπου η Κομισιόν έχει δημοσιοποιήσει τις προ σπάθειες της και χρειάστηκε να αναφέρω στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι ο στόχος είναι να μειωθεί το ρίσκο συνολικά. Έχουμε συμφωνήσει ότι αυτή η μείωση του κινδύνου πρέπει να συνοδευτεί από έναν επιμερισμό του κινδύνου. και έχει ασκηθεί κριτική σε ορισμένες χώρες, κρατημέλη, τα, οι οποίες ε, θεωρείται ότι έχουν μπλοκάρει αυτόν τον επιμερισμό του κινδύνου. Και υπάρχουν κατηγορίες, ε, λόγω κατηγορίες. Και εύλογο είναι όταν κανείς ε, ακούει τέτοιου τύπου κατηγορίε να προσπαθεί να υπεραμεινθεί τι θέσει του γιατί πράγματι όπω είπατε το ζήτημα του Έντι έχει ε, συζητηθεί επί μακρόν και συνδέεται με την ολοκλήρωση τη αρχιτεκτονική τη Τραπεζικής Ένωση. Και θα έλεγα ότι μάλλον τις απαντήσεις θα μας δώσουν τα αποτελέσματα των εκλογικών αναμετρήσεων την επόμενη χρονιά. Χαίρομαι που έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις στο τραπέζι πάντως αυτή τη στιγμή, έτσι ώστε η επερχόμενη Προεδρία της Μάλτας να ξεκινήσει τη συζήτηση και να καταλήξουν σε συμφωνίες. Ε, όπως σας είπα όμως, η τεχνική συζήτηση θα ξεκινήσει ήδη από αύριο. Δεν βλέπω κανένα λόγο να καθυστερήσει η συζήτηση για το έντις. Και εξάλλου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πει ότι θα χρειαστεί χρόνο για να καταλήξει σε μια κοινή θέση. Ε, στην συζήτηση την χθεσινή για τα ενημερωτικά δελτία, για την οδηγία προσπέκτους, ε, συναντήθηκα με συναδέλφου σας και μου είπαν ότι το θέμα αυτό θα συζητηθεί στο, στο Στρασβούργο. Θα υπάρξει μια συζήτηση γιατί υπάρχουν πολύ διαφορετικές απόψεις μεταξύ των Ευρωβουλευτών. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο συνδέεται και συνδυάζει παλαιότερους και σημαντικούς στόχους, αλλά επίσης και θέματα που ε, έχει θεωρηθεί ότι έχουν συζητηθεί και κλείσει στο παρελθόν. Το σίγουρο είναι ότι κατά την άποψή μου δεν θα καταφέρουμε να υπάρξει μια αμοιβεοποίηση του κινδύνου και των εγγυήσεων για τον κινδύνο στο ευρωπαϊκό ε, τραπεζικό σύστημα, εάν πρώτα δεν καταφέρουμε να συμφωνήσουμε στον τρόπο με τον οποίο στο τραπεζικό σύστημα κάθε χώρας θα μειωθεί ο κίνδυνος. Γιατί υπάρχουν ορισμένες χώρες στις οποίες μπορεί να υπάρξουν προβλήματα. Και επίσης, ε, κλείνοντας την παρέμβαση μου για το θέμα αυτό. Ε, πιστεύω ότι η τεχνική ανάγνωση του κειμένου κατάρθρο ήταν ε, σωστό που έγινε στο Συμβούλιο, ένα σκόπιμο που έγινε στο Συμβούλιο, γιατί μπορέσαμε να μπούμε στις λεπτομέρειες και να καταλάβουμε ακριβώς τι προτείνεται. Thank Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Μπερές, η επόμενη μιλητρία Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Δεν θα ήθελα να επανέλθω σε παλαιότερες συζητήσεις, αλλά έχω την εντύπωση ότι ε, πραγματικά επιμένουμε στη μείωση του κινδύνου για να μην συζητήσουμε τον επιμερισμό. Αλλά, τέλος πάντων, εγώ θα σταθώ περισσότερο στο, στη διάσταση της μακροοικονομικής σταθερότητας που αναφέρατε και το Κοινοβούλιο έχει εκφράσει την βούλησή του στον τομέα αυτών. Ε, επικυρώνοντας το ότι, ε, μάλλον λέγοντας ότι δεν θα έπρεπε να επιβληθούν πρόστιμα στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Πιστεύω ότι αυτή η απόφαση ήταν σοφή, γιατί αυτές οι δύο χώρες έχουν παρουσιάσει και ξεκινήσει να εφαρμόζουν ορθά μέτρα για να ε, ισοσκελίσουν τους προπολογισμούς τους. Αλλά επίσης δεν θα πρέπει να τεθεί και το ζήτημα του κυκλικού χαρακτήρα, του προστίμου και της ε, μη χρήση των τριαρθρωτικών ταμείων που οδηγεί σε ύφεση αυτή. Επομένως, δεν θα πρέπει να ξαναδούμε ουσιαστικά και εκθεμελίων αυτήν την πολιτική. Και εσείς τι πιστεύετε γι' αυτό. Εγώ θα έλεγα ότι το ζήτημα μπορούμε να το δούμε ως ε, το τι κάναμε μετά την έκθεση των πέντε προέδρων. Δυστυχώς δεν υπήρξε η απαιτούμενη πρόοδος και δυστυχώς διαπίστωσα ότι και στην ε, Σύνοδο Κορυφής της Πρατισλάβα ε, δώσαμε μεγαλύτερη έμφαση στην ασφάλεια και στην άμυνα εις βάρος της ε, σημασίας που θα έπρεπε να δίνουμε στην ανάπτυξη. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μας λέει όλο και πιο συχνά, όλο και μεγαλύτερη επιμονή ότι χρειάζεται να βελτιώσουμε την ε, ε, χρηματοοικονομική κατάσταση της ζώνης του ευρώ. Χωρίς μικρόφωνο, δεν ακούνε οι διερμηνείς. Πρέπει να φύγω σε πέντε λεπτά. Έχω μια αντιλημμένη υποχρέωση και πρέπει να φύγω σε πέντε λεπτά. Θα μπορούσα μήπω να κάνω τώρα την ερώτησή μου πριν να απαντήσει ο Υπουργό. Uh, uh, τώρα δεν συνηθίζεται αυτό. Θα έπρεπε να μας είχατε ενημερώσει. Τώρα εντάξει θα δώσω το λόγο στον Υπουργό για να απαντήσει και μετά θα σας δώσω χρόνο. Ε, ε, ε, λοιπόν, θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλα τα θέματα μαζί. Ε, όσον αφορά την Ευρωζώνη, πρέπει να σας πω ότι έχουμε επιτύχει συνένεση ε, επί του γεγονότος ότι τα φορολογικά εισδήματα θα πρέπει ε, να τα αντιμετωπίσουμε με διαφορετικό τρόπο. Εν πάση περιπτώσει, ε, οπωσδήποτε θα πρέπει να δείξουμε για ορισμένα θέματα θάρρος, έτσι ώστε να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Υπάρχουν πολλές προτάσεις όσον αφορά την ε, ε, διασφάλιση ε, για τον έλεγχο της ανεργίας. Υπάρχουν πάρα πολλές προτάσεις. Κοιτάξτε, εμείς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να πούμε ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η νομισματική ένωση, η αρχιτεκτονική της ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, η πραγματικότητα είναι αυτή που είναι ε, και το περιβάλλον δεν είναι το καλύτερο δυνατό ε, είπα και στην αρχή ότι περιμένουμε και πρέπει να περιμένουμε τα αποτελέσματα αυτών των μεγάλων εκλογικών αναμετρήσεων της επόμενης χρονιάς και επομένως ε, καταλαβαίνετε ότι πολλά πράγματα μπορεί να αλλάξουν. Ακόμα δεν μπορούμε να πάρουμε τελική θέση απέναντι σε όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία ε, ανέφερα στην εισήγησή μου την αρχική, βλέποντας και το παράδειγμα της Ισπανίας και της ε, Πορτογαλίας. Ναι, όντως ε, μπορεί να είμαστε λίγο με την πλάτη στον τοίχο σε ορισμένε περιπτώσεις, αλλά οδοί υπάρχουν έτσι ώστε να εξελιχθούμε. Τώρα, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι αν δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τους κανόνες, να τους αλλάξουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Σταπάκη. Κύριε Υπουργέ, σε ό,τι αφορά την Αμισματική Ένωση, είπατε ότι χρειάζεται περισσότερη δράση. More action is needed, πράγματι. Δεν είναι καλές η, καλή εικόνα. Εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητούμε συνέχεια τις πολιτικές, ποιες είναι καλές για και κατάλληλες για την Ευρωζώνη, για να υπάρξει ανάπτυξη. Υπάρχουν δύο ρεύματα. Η μία σχολή λέει ότι δεν μπορούμε στο μέλλον να συσσωρεύουμε χρέος, αυτό θα πει πολιτική λιτότητα και η δεύτερη λέει ότι θέλουμε περισσότερο περιθώριο για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι και οι απόψεις αυτές ε, αλληλοσυγκρούονται σε όλες τις συζητήσεις που έχουμε εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο. Το δεύτερο είναι αυτό που είπατε ότι σίγουρα χρειαζόμαστε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Αυτό είναι σαφές θα πρέπει να υπάρξει εξηγένση δημοσιονομική. Χρειάζονται δημοσιονομικές, συγγνώμη, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και σε ό,τι αφορά τι κοινωνικέ παροχέ, φορολογία κτλ. Όλα αυτά είναι απαραίτητα. Εσείς είστε προεδρεύων τώρα ε, στο ε, Συμβούλιο Κοφίν και σας ερωτώ υπό αυτήν την ιδιότητα η αλλαγή δομών ε, μέσα στον προπλασμό είναι κάτι που έχει αναφερθεί ή απλά λέμε κάνουμε το τάδε, κάνουμε το δίνα. Συγκεκριμένα έχει συζητηθεί το πώς τα μεμονωμένα κράτη-μέλη θα πρέπει να γίνουν ε, μεταρρυθμίσεις. Τι μεταρρυθμίσεις διεθνωτικές πρέπει να γίνουν συγκεκριμένα σε κάθε κράτος μέλος. Ε, ε, Κοιτάξτε, Πρέπει να σας πω ότι το ζήτημα σήμερα είναι η Ευρωζώνη και το λέω με μεγάλη ευγένεια και εγώ ως πρόεδρος προεδρεύων του ΕΚΟΦΗΝ δεν ε, ε, ήρθα εδώ για να μιλήσω για τον προϋπολογισμό. Εν πάση περιπτώσει, ε, είναι αλήθεια ότι ξεπερνάμε λίγο, προχωράμε πέρα από το νομοθετικό πλαίσιο. Επαναλαμβάνω, επαναλαμβάνω ότι η ε, Κομισιόν ε, έχει έχει κάποιες συστάσεις όσον αφορά το δημοσιονομικό ε, πλαίσιο και όσον αφορά μέτρα τα οποία θα πρέπει περαιτέρω να ληφθούν από το Eurogroup ε, και ε, αυτά βρέθηκαν μη συμβατά με τους ισχύοντες κανόνες το ας πούμε το σύμφωνο για την σταθερότητα και την ανάπτυξη δεν περιέχει τέτοιους κανόνες και επομένως θα πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε κάποια λύση πέρα από αυτούς τους ε, κανόνες. Δηλαδή προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν ε, ε, στο Eurogroup. Συζητούμε και για οριζόντιες πολιτικές, ας πούμε, ε, τις δαπάνες των κρατών μελών, ε, ας πούμε διαδοτικέ ε, αλλαγές όσον αφορά το τμήμα των δαπανών κλπ. Θυμάμαι ας πούμε ε, ότι έγινε μια παρουσίαση από τον συνάδελφο Παντοάν ε, σχετικά με την ε, κατάσταση στην Ιταλία και ο αντίστοιχος υπουργό της Ισπανίας για τις δαπάνες της Ισπανίας αλλά μιλάμε πάντα για το Eurogroup, τα προβλήματά του και την ανάκτηση αυτών των προβλημάτων. Προσπαθούμε να βρούμε νέες πρακτικές οι οποίες θα μας βοηθήσουν να ξεπεράσουμε τα προβλήματα και πάντα όσον αφορά τους κανόνες που έχουν περάσει ε, την νομοθετική διαδικασία, το 2 το 6-pack, ε, το σύμφωνο σταθερότητας. Ε, κοιτάξτε, και επίσης έχουμε και το νέο εργαλείο το οποίο αφορά την απλούστευση των κανόνων Ε, υπάρχουν ακόμα πολλά τεχνικά ζητήματα τα οποία μπορεί να έχουν ε, άμεσο αντίκτυπο ε, στις δημοσιονομικές πολιτικές. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Ε, εντάξει, δεν λέτε ότι, είναι, ότι το, η προτάση fiscal stand για τη, της Κομισιόν ε, δεν είναι νομιμοποιημένες. Απλώς ο τρόπος με τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί αυτό το fiscal stand είναι λίγο διαφορετικός. Συνάδελφος Γεζέκ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ για την ε, προσέγγιση σας ε, και για τον τρόπο με τον οποίο ε, μας δίνετε την δυνατότητα, μας δώσατε μάλλον τη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε αυτή τη συμφωνία για τα προσπέκτους πριν από 12 ώρες. Εγώ είμαι εισηγητής και βρισκιώδη σε, σε σχετικά ζητήματα και να σας πω ότι εξ όσων γνωρίζω φαίνεται ότι δεν υπάρχει μεγάλη διάθεση ε, για πολύ μεγαλύτερη διαφάνεια, κυρίως όσον αφορά ε, το μητρό των beneficiary, beneficiary owners. Ε, η διαφάνεια όμως είναι σημείο κλειδί ε, για μας ε, έτσι ώστε ε, να καταφέρουμε να καταπολεμήσουμε την απάτη. Και καταλαβαίνετε ότι στην περίπτωση πραγματικών δικαιούχων η διαφάνεια μετράει πάρα πολύ. Δεύτερο, τι θα κάνει γι' αυτό λοιπόν η Κομισιόν. Δεύτερο ε, που με απασχολεί αφορά την Σλοβακική Προεδρία. Πιστεύουμε ότι ήταν πολύ επιτυχημένη, κυρίως ε, ε, για μια χώρα σχετικά νέα. Ωστόσο, ποια είναι τα στοιχεία τα οποία θεωρείτε κλειδιά ε, όσον αφορά το δικό σας πλαίσιο αρμοδιοτήτων. Ποια θα θεωρούσατε ε, επιτυχημένα στοιχεία και βήματα για το μέλλον. Επίσης, ε, και τελειώνω, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την επιτυχή Σλοβακική Προεδρία. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ ε, για τα καλά σας λόγια. Ίσως ε, να ξεκινήσω ε, με την ερώτηση που μου κάνατε, δηλαδή τι θα θεωρούσα σημαντικό στοιχείο για, τις, για την επόμενη περίοδο. Ίσως ίσως θα έλεγα να προωθήσουν το τις 2 που είναι σχεδόν έτοιμο. Ε, είχαμε και μία διάσκεψη στο Παρίσι, τα διάσκεψη του ε, ΟΣΑ Ε, όπου ήταν παρόντες ε, πολύ σημαντικοί εκπρόσωποι της μάχης κατά της ε, φοροδιαφυγής και ήταν παρούσα και η επερχόμενη Μαλτέζικη Προεδρία. Βεβαίως η Μάλτα δεν είναι και κύριος παίκτης όσον αφορά το θέμα αυτό, αλλά παρόλα αυτά σε μία περίοδο πολιτικής αναταραχής. Ε, αυτό που θα έλεγα στους συναδέλφους από την ε, Μάλτα ε, είναι να ξεχάσουν τι λένε τα μέσα ενημέρωσης, να μην τα ακούνε και πάρα πολύ και να εστιάσουν στην, στα θέματα που είναι σημαντικά. Και το σημαντικό είναι να συνεχίσει η προσπάθεια και η δουλειά για την Τραπεζική Ένωση επίσης την ε, μείωση ε, κινδύνου με συγκεκριμένα στοιχεία καθώς επίσης και συνέχιση των τριμερών διαλόγων όσον αφορά την τιτλοποίηση ας πούμε. Αυτά είναι σημαντικά θέματα και όλοι μας ανυπόμονα περιμένουμε τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής καθώς επίσης και την αξιολόγηση των πέντε προηγουμένων εκθέσεων όσον αφορά την Νομισματική Ένωση, όσον αφορά την ε, πρωτοβουλία για το ξέπλυμα χρήματος. Ε, αυτή είναι συνολική πρωτοβουλία, πάρα πολύ σημαντική. Δύο φορές έχω αντιμετωπίσει το ε, θέμα αυτό το δημοσιοποιήσαμε και το κάναμε επίτηδες ε, γιατί θεωρούμε ότι μια και πρόκειται για μια δημόσια πληγή, ε, για μια δημόσια ε, κατάσταση θα πρέπει να δημοσιοποιούνται κάποια στοιχεία. Πρέπει να γίνει μια έκκληση σε δημόσιο επίπεδο αν θέλετε. Πρέπει να προχωρήσουμε το θέμα αυτό, έστω και αυτές τις δέκα μέρες που μας ε, μένουν και βεβαίως ε, και οι υπόλοιποι θα συνεχίσουν. Ε, δεν θέλω να μπω σε άλλες λεπτομέρειες γιατί καμιά φορά η υπερβολική δημοσιοποίηση στοιχείων δυναμητίζει την επιτυχία αλλά ξέρετε ότι έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ και όσον αφορά και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και επίσης στην ανάκτηση χρημάτων τα οποία αν τα είχαμε στη διάθεσή μας θα μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε με πολύ καλό τρόπο. Ε, επομένως, ε, να εύχεστε να προχωρήσουμε όσο γίνεται περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ. Thank Δημήτρης Παπαδημούλης. Ευχαριστώ, Δημήτρης Παπαδημούλης. Mr. you can use your headphones. Μπορείτε να βάλετε τα ακουστικά σας, κύριε Κάζιμιρ, γιατί δεν έχετε φαντάσμα ακόμη μάθει καλά ελληνικά μέχρι να μάθετε και ελπίζω να μάθετε. Πιστεύω ότι η Σλοβακική Προεδρία ήταν μια παραγωγική Προεδρία και θεωρώ καλά νέα για την Ελλάδα το γεγονός ότι δεν αναφερθήκατε ε, στην ελληνική οικονομία στην εισαγωγική σας ομιλία γιατί από ό,τι είδα και από τις ανακοινώσεις και του Eurogroup και του ECOFIN και της Κομισιόν ελληνική οικονομία σημειώνει επιδόσεις καλύτερες από τις προβλέψεις που υπήρχαν για τα έτη 15 και 16 και ελπίζω να συμβάλλετε ως μέλος του ΕΚΟΦΗΝ και μετά την ολοκλήρωση της Προεδρίας έτσι ώστε να ολοκληρωθεί σύντομα η δεύτερη αξιολόγηση και να μπει σε έναν ενάρετο κύκλο ανάπτυξης η οικονομία της χώρας μου. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πολύ σύντομα δύο πράγματα κύριε Κάζιμερ. Το πρώτο, στην ατζέντα της Σλοβακικής Προεδρίας που μας παρουσιάσατε πριν λίγους μήνες ήταν το Banking Union. Πριν λίγες ημέρες εδώ ο Μάριο Ντράγκη μας είπε ότι δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η τραπεζική ενοποίηση χωρίς τη δημιουργία του τρίτου πυλώνα, του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εγγύησης Καταθέσεων. Και ότι η ασάφεια και η αστάθεια, η διεθνής, επιβάλλει την θωράκιση της τραπεζικής ένωσης και με τον τρίτο πυλώνα, γιατί χωρίς τρίτο πυλώνα δεν υπάρχει τραπεζική ένωση θα ήθελα να σας ρωτήσω αν συμμερίζεστε την άποψη Ντράγκη για το ΙΔΙΣ και δεύτερον τι σκητάλη παραδίδεται στην Προεδρία της Μάλτας σε ό,τι αφορά την πρόοδο σε αυτό το φάκελο που είχε ξεκινήσει και από την προηγούμενη Προεδρία την Ολλανδική. Και το δεύτερο, τον Ιούλιο του 2016 το Συμβούλιο κατέληξε σε κάποιες συστάσεις προς τη Γερμανία για τις μακροοικονομικές ισορροπίες που, ανισορροπίες που παρουσιάζει με υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, ζητώντας αύξηση των δημόσιων επενδύσεων και τόνωση ιδιαίτερα των χαμηλών εισοδημάτων προκειμένου να μπορούν ευκολότερα να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Θα ήθελα να μου πείτε από τον Ιούλιο μέχρι τώρα αν έχετε προχωρήσει σε αξιολόγηση αυτών των μέτρων δεδομένου ότι στην ίδια εκτίμηση και στις ίδιες συστάσεις για μακροοικονομικές ισορροπίες στη Γερμανία που βλάπτουν και την συνολική ευρωπαϊκή οικονομία έχει καταλήξει και η Κομισιόν. Και επειδή τα ελλείμματα του Νότου και τα πλεονάσματα του Βορρά αλληλοτροφοδοτούνται, θα ήθελα να μου πείτε εσείς που είστε στο κέντρο της Ευρώπης πώς βλέπετε αυτή την εξέλιξη. Hovorili ste o nevyhnutnosti e, dokončiť Μιλήσατε e, για την Τραπεζική Ένωση που πρέπει να ολοκληρωθεί, είπατε. Και εγώ ρωτώ τι είναι τελικά πιο σημαντικό μια ατελής νομισματική ένωση, μια ατελής τραπεζική ένωση. Αυτή τη στιγμή η Τραπεζική Ένωση δεν είναι ολοκληρωμένη. Αυτά τα θέματα όμως θα μπορούσαμε να τα θεωρήσουμε συγκρίσιμα μεταξύ τους. Και μιλώντας ανοιχτά και ειλικρινά σε τεχνικό επίπεδο, και επειδή όπου να είναι τελειώνει η Προεδρία μας και έρχεται ε, η Μαλτέζικη Προεδρία, ουσιαστικά προσπαθούμε να ανακτήσουμε το χαμένο έδαφος, γιατί περιμέναμε μήνες στις προτάσεις της Κομισιόν. Και πραγματικά δεν νομίζω ότι πριν ολοκληρωθεί ο κύκλος των εκλογών ε, του χρόνου θα μπορέσουμε να έχουμε ε, κάνει μεγάλες τομές και να έχουμε προχωρήσει σημαντικά σε αυτά τα μέτωπα. Και επειδή όπου να είναι κατέρχομαι από το αξίωμα του προεδρεύοντα του ΕΚΟΦΗΝ, μπορώ να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας. Ε, νομισματική Ένωση ή Τραπεζική Ένωση ε, τόσο ρηξικέλευτες πρόοδους ολοκλήρωση αυτών των θεμάτων να μην τα περιμένουμε του χρόνου. Δεν ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση, υπάρχει προθυμία για να βοηθήσουμε και εμείς ε, την επόμενη Προεδρία. Απλά πρέπει να βλέπουμε την πραγματικότητα. Έχουμε αυτές τις εκλογές του χρόνου, θα επηρεάσουν. Μίλησετε για την Ελλάδα. Γνωρίζετε. Και αν το πω και εγώ, ε, είναι σημαντική πληροφορία ίσως για εσάς, ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα και ο κ. Τσακαλώτος συγκεκριμένα ως Υπουργός Οικονομικών έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο. Είναι εξαίρετος ο Υπουργός Οικονομικών της χώρας σας και χέρι της αμέριστης εμπιστοσύνης των συναδέλφων του, γιατί αν δεν την είχε δεν θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε αυτό το project, διότι φυσικά πρέπει να ακολουθείται μια κοινή προσέγγιση από όλου. Και τις τελευταίες ημέρες αυτό που μας απασχόλησε είναι για παράδειγμα σε ποιο βαθμό θα πρέπει να υπάρξει μια μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας. με στόχο ε, η χώρα να ε, προσεγγίσει όσο το δυνατόν περισσότερο τα βέλτιστα ευρωπαϊκά πρότυπα. Μιλάμε για εργασία, για αγορά εργασία. Δεν είναι δική μου βέβαια αρμοδιότητα, ούτε δική μου ειδικότητα. Πάντω, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολύ καλά νέα για την Ελλάδα και για την Ευρωζώνη εγκρίθηκαν αυτά τα βραχυπρόθεσμα μέτρα και καταφέραμε αυτή τη συμφωνία να την ολοκληρώσουμε. και σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Δηλαδή έχουμε προχωρήσει ακριβώς όπως είχαμε συμφωνήσει. Thank you, Darius Rosati. Yes, thank you, Chairman, and uh, thank you, Minister, for being. Σας ευχαριστώ, Κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ τον Υπουργό της Σλοβακίας για την παρουσία του εδώ. Η πρώτη μου ερώτηση αφορά τις μεταρρυθμίσεις με στόχο την αύξηση της ανθεκτικότητας της Ευρωζώνης. Έχουμε ασχοληθεί με την χρηματοδοτική ικανό... δημοσιονομική ικανότητα της Ευρωζώνης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αναρωτιέμαι Ποιε είναι οι αντίστοιχε συζητήσει που έχουν γίνει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Είναι σε αρχικό στάδιο ή αν έχει προχωρήσει περισσότερο η συζήτηση ε, αυτή. Το δεύτερο ερώτημά μου αφορά στον φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Πριν από πέντε χρόνια η Επιτροπή υπέβαλε την αρχική της πρόταση και από τότε δεν έχει σημειωθεί και μεγάλη πρόοδο στον τομέα αυτών. Θα έλεγα ότι ο αρχαιοκός ενθουσιασμός έχει πλέον χαθεί. Τουλάχιστον από ο ενθουσιασμός που είχαν επιδείξει κάποια κράτη-μέλη. Επομένως το ερώτημά μου είναι ε, η πρωτοβουλία αυτή συνεχίζει να είναι εν ζωή. Και αν όχι, ποια είναι τα σημαντικότερα εμπόδια ε, που σταματούν την πρόοδο. Začnem, začnem odpovedou v oblasti FTT. A... Σε ό,τι αφορά το φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, η χώρα μου είναι μεταξύ των χωρών που έχει ενισχυμένη συνεργασία, αλλά εγώ αυτή τη στιγμή ομιλώ από την ιδιότητα του πρόεδρου του ΕΚΟΦΗΝ. Μαζί με Πορτογάλους εμπειρογνώμονες καταφέραμε, και παρότι μπορεί να μην φαίνεται προς τα έξω, καταφέραμε πολλά σε ό,τι αφορά τα βασικά στοιχεία της συμφωνίας. Και οι Αυστριακοί μιλούν για μια ευρεία βάση και για χαμηλούς συντελεστέ. Αυτή είναι η αρχή. Και από αυτόν συμφωνήσαμε μόνο μέχρι τώρα. Και Επίση συμφωνήσαμε να υπάρχει ένας ελάχιστος αριθμό εξαιρέσεων. Αυτοί, αυτοί είναι οι βασικοί άξονε. Αυτέ ε, είναι οι αρχές. Σε ό,τι αφορά τώρα αυτή τη ε, συνεργασία είναι κάτι που είναι γνωστό σε όλους. Και σε ό,τι αφορά αυτή τη συνεργασία και αυτή τη φορολογία λέμε ότι αυτό θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο γενικό και σφαιρικό. Ο Βόλφκαν Κασόιμπλε, ο Γερμανός υπουργό Οικονομικών, υποσχέθηκε ότι όταν θα επειδή έχουν την προεδρία του G20, η Γερμανία θα προσπαθήσει να την αξιοποιήσει για να προχωρήσει. Και αυτό το θέμα βέβαια δεν υπάρχει πίεση, δεν ε, δεχόμαστε από κανένα πίεση για την ενισχυμένη αυτή συνεργασία. Εξάλλου είναι ζήτημα ομοφωνία γιατί πρόκειται για θέμα άμεσης φορολογίας. Πρέπει να προστατεύσουμε αυτά τα σχέδια και προγράμματα που μπορούν να ε, δρομολογήσουν ε, οικονομική ανάπτυξη. Απλά υπάρχουν κάποια θέματα που αρχίζουν να παρισφρίουν σε άλλα και επηρεάζουν. Το θέμα είναι να προχωρήσουμε. Δεν πέθανε λοιπόν ο φόρος των ψηφιακών συναλλαγών. Υπάρχουν 10 κράτη-μέλη Συνεχίζει η δουλειά, Συνεχίζει δουλειά μας πάνω σε αυτό, αλλά θα πρέπει να το δούμε πιο πολύ ως οικονομικό και όχι τόσο ως πολιτικό σχέδιο. Μιλήσατε για τη μουσομική ικανότητα της Ευρωζώνης. Είναι ένα θέμα, το ανέφερε και η κύρα Μπερές, για την ε, ολοκλήρωση της αρχιτεκτονικής της ε, ενός κεφαλαίου αγορών. Έχουμε και το πακέτο Juncker. Το FC2 ήθελε, ε, απαιτούσε αυτή την δημοσιονομική ικανότητα για να μπορεί να τα αποκριθεί η Ευρωζώνη σε κραδασμούς, που είναι ένα θέμα ταμπού βέβαια αυτή την ίδια δημοσιονομική ικανότητα. Είναι κάτι που πολλέ χώρε δεν θέλουν να εφαρμόσω. Επειδή όμως έχω αυτή την ελευθερία τώρα να μιλάω πιο ανοιχτά, θα ήθελα να λέμε στο μέλλον ότι το ΕΦΣΥ ήταν ένα είδος ε, δημοσιονομική ε, ικανότητα σε εμβριακή κατάσταση και δεν θα έπρεπε να ταφεί αυτή η προσπάθεια πολλοί αρνήθηκαν να συζητήσουν αυτό το θέμα. Αλλά το να στηρίξουν το ΕΦΣΥ ε, τους δίνει καθαρή συνείδηση για να δουν τι θα κάνουν μετά και αν θα συνεχίσουν ή δεν θα συνεχίσουν με την ολοκλήρωση της αρχιτεκτονικής της ΟΝΕ. Thank you. Σας ευχαριστώ. Κύριε ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, όπως είπατε πολλά έγιναν όσον αφορά ε, την, ε, τα δημοσιονομικά. Ξέρετε ότι το Κοινοβούλιο έχει δουλέψει πάρα πολύ έτσι ώστε να σταματήσουν πλέον αυτή η φορολογική ε, παράδειση ε, καθώς επίσης και οι ειδικέ συμφωνίες. Αλλά είδαμε ότι έχουν ε, μεταξύ του 2013 και του 2015 έχουν τριπλασιαστεί οι αριθμοί των ειδικών φορολογικών ε, συμφωνιών. Επομένως ε, θα πρέπει να σταματήσει αυτή ε, η κατάσταση, αλλά διαπιστώνω ότι υπάρχουν κάποιοι δισταγμοί. Μπορείτε να μας πείτε ποιες είναι οι χώρες οι οποίες διστάζουν περισσότερο. Εγώ είμαι απολύτως πεπισμένος ότι όσο δεν υπάρχουν ή δεν προβλέπονται κυρώσεις και όσο δεν υπάρχει πλήρης διαφάνεια δεν πρόκειται να ε, βελτιωθεί η κατάσταση. Επίσης όσον αφορά Επίσης ε, υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που λένε ότι δεν ε, θα μπορέσουμε ε, να λύσουμε το θέμα της πραγματικής διαφάνειας και το θέμα της πραγματικής τραπεζικής ένωσης μόνο μέσω της λύσης ορισμένων προβλημάτων που σχετίζονται με την Ένωση των Κεφαλαίων Αγορών. Είσαστε της ιδίας απόψεως και τι μπορείτε να μας πείτε πάνω σε αυτό. Ja chcem povedať, eh, Κοιτάξτε, εγώ έρχομαι από μια χώρα όπου η αποτελεσματικότητα ε, της ε, ε, της, φορολογίας ε, έχει τροποποιηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και πρέπει να σας πω ότι αναγκαστήκαμε στην ουσία να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό, γιατί και λόγω της εξυγίανσης ε, τα δημόσια οικονομικά είναι συγκεκριμένα και ε, βεβαίως ε, η δυνατότητα να υπάρξει πρωτογενές πλεόνασμα και η υποχρέωση του κράτους να επενδύσει στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής ήταν πολύ σημαντικά θέματα. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς σε αυτό επικεντρωθήκαμε. Πιστεύω ακράδαντα ότι ένα από τα ευτυχή στοιχεία της ε, κρίσης ε, ήταν ότι έχει αλλάξει η γενική προσέγγιση όσον αφορά την φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή. Ε, ε μάλιστα επιβράβευσα τον ε, σαν Κούριο όσον αφορά τα όσα ε, ε, επέτυχε στον αγώνα κατά της φοροδιαφυγής. Για πολλές δεκαετίες λέγαμε απλώς ότι το σύστημα πρέπει να αλλάξει και φυσικά η αλλαγή δεν μπορεί να προέλθει από τη μια στιγμή στην άλλη. Ε, οι αλλαγέ όμως τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ μεγάλες. Αν δει κανεί τη δεκαετία του 70, τη δεκαετία του 80, η Συνολική Συμφωνία για την Ανταλλαγή ε, ε, πληροφοριών ήταν σε εμβριακό στάδιο ενώ τώρα βρισκόμαστε ε, πρώτων θυρών της εφαρμογής της ανταλλαγής πληροφοριών και βλέπουμε ότι αρχίζει πανικός στους φορο διαφεύγονται σε ανθρώπους που για δεκαετίες δεν είχαν πληρώσει φόρους. Επομένως, καταλαβαίνω ότι θα πρέπει να κρατήσουμε αυτήν την ε, καλή πορεία. Ε, κάποιες επικρίσεις ε, βέβαια σχετίζονται ίσως με το ότι δεν προχωρήσαμε αρκετά ακριβά. Εν πάση περιπτώσει, όσον αφορά το ε, υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία δεν καταλαβαίνουν ε, οι πολίτες ε, και δεν τα αντιμετωπίζουν σωστά και τα μέσα ενημέρωσης. Ε, ξέρουμε ότι υπάρχουν λόμπι τα οποία προσπαθούν να περάσουν τους δικούς τους κανόνες και από την άλλη πλευρά γνωρίζουμε ότι υπάρχουν δισεκατομμύρια τα οποία χάνουν τα κράτη-μέλη μέσα από τα χέρια τους. για πολλούς και διάφορους λόγους. Γι' αυτό λοιπόν η Κομισιόν ε, ε, ξεκίνησε ε, ακριβώς ε, διάφορες διαδικασίες επί παραβάση συγκεκριμένα για μη εφαρμογή των όρων του ανταγωνισμού και υποχρεώνοντας τα κράτη να παράσχουν οριζόντιες πληροφορίες σχετικά με παραβάσεις ας πούμε των κανόνων για κρατικές επιδοτήσεις ζητούμε ε, οριζόντιες ε, πληροφορίες. Ε, επομένως, θέλω να σας πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ για τον βαθμό συνεργασίας που έχουμε με την Κομισιόν και με την Ταξίδ και ε, Βεβαίω, ε, ε, θα ήθελα εδώ να πω πόσο σημαντικό είναι και ο ρόλος, ο υποβοηθητικό ρόλος και του ΩΣΑ και του G20. Οι χώρες του G20 παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και δεν θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε χωρίς την υποστήριξη των χωρών του G20. το θέμα της κοινή φορολογικής βάσης ανακοινήθηκε και προωθήθηκε και από την δική μας ε, Προεδρία. Και αναζωογονήθηκε κατά κάποιο τρόπο. Εάν δει κανείς ε, πώς ε, ξεκίνησε το θέμα της κοινή φορολογικής ε, βάσης ε, μπορεί να καταλάβει πόσο έχει αλλάξει το υπόδειγμα. Βεβαίως απαιτήθηκε πάρα πολύ δουλειά, αλλά χρειάζεται ακόμα πολύ δουλειά. Πάντως έχουν αλλάξει οι νοοτροπίες προς το καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ. Ο Μπερτ Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα και εγώ να συνεχίσω πάνω σε αυτό που εσείς είπατε τελευταίο για το φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ε, και τη φορολογική βάση, την ενωπημένη. Έχουμε όμως και άλλα θέματα που μπλοκάρουν τα κράτη ε, παραδείγματο χάρη, σε ό,τι αφορά το φόρο προστέμενη αξία. Ε, έχουμε το δεκαετία του 90 αυτό το σύστημα για το ΦΠΑ ε, και έχουμε 160 δι ε, τρύπα στα έσοδα, στα φορολογικά. Τι έχει γίνει τα 23 τελευταία χρόνια, σχεδόν τίποτα. Αποφασίζουμε συνέχεια ότι θα έχουμε καλύτερη συνεργασία και τελικά δεν γίνεται τίποτα. Μένουμε στα λόγια, μένουμε σε δηλώσεις από το ΕΚΟΦΗΝ, από τα κράτη-μέλη και από την Κομισιόν. Και επομένως ε, το ερώτημά μου είναι πώς θα καταφέρουμε στην προκειμένη περίπτωση μεταρρύθμιση του ΦΠΑ, ε, γιατί υπάρχει και ε, συγκεκριμένο άρθρο της συνθήκης ε, που μας ε, επιτάσσει να προχωρήσουμε σε αυτή την μεταρρύθμιση. Έχουμε το, τους Αυστριακούς, τους Τσέχους. Θα μπορούσαμε τα παραδείγματά τους να τα ακολουθήσουμε σε ένα είδος πιλωτικού προγράμματος. Ποιο θα είναι το επόμενο βήμα λοιπόν και η επόμενη ερώτηση είναι έχουμε την Εξεταστική Επιτροπή Πάνα για τα έγγραφα του Παναμά. Και εκεί υπάρχει και το ξέβλημα χρήματο και σχετική οδηγία, Ευρωπαϊκή Αγγελία και αρμοδιότητε. Από ό,τι ξέρω, συμφώνησε και το ΕΚΟΦΗΝ ε, για ε, αφορολογική απάτη πάνω από 10 εκατομμύρια είναι ευρωπαϊκή αρμοδιότητα. Αλλά και εκεί υπάρχει εμπλοκή για τα θέματα ξεπλήματος ε, χρήματος. Όπου κοιτάμε λοιπόν για τα φορολογικά ζητήματα, βλέπουμε να μπλοκάρουν την κατάσταση τα κράτη-μέλη. Εμεί θέλουμε να υπάρχει φορολογική δικαιοσύνη. Αυτή είναι κεντρικό είναι κεντρικός πυλώνας ε, για την περαιτέρω εξέλιξη της Ευρώπης. Ε, δεν μπορούμε ούτε την Amazon ούτε την Apple να αφήνουμε να τα διαγράφουν όλα, να, τα, ε, να κάνουν ό,τι θέλουν. Ακούσαμε να λέγεται για την Apple ε, στην Ιρλανδία. Ο Ιρλανδό Υπουργό ε, Οικονομικών ήρθε και μα είπε ότι ακολουθούμε τι ίδιε περιγραφέ και κανόνε με την Apple και ό,τι, όπως με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία. Μα είπατε εσεί ε, τον απολογισμό τη Προεδρία, μα μιλήσατε για την Μαλτέζικη Προεδρία. Τι περιμένετε από τη Μαλτέζικη και από την Εστονική Προεδρία, που είναι οι επόμενε δύο, το 2017. Poznáte temu daňovej suverenity. A viete, že e, v niektorých krajinách... Για το ζήτημα της φορολογίας. Όλοι γνωρίζετε την θέση χωρών και κυβερνήσεων που επιμένουν ιδιαίτερα στο ζήτημα της κυριαρχίας, της, της δυνατότητας κάθε κράτους να ορίζει το φορολογικό του σύστημα. Έχουν ξεκινήσει ακόμα και πρωτοβουλίας για να προστατευτεί αυτή η φορολογική κυριαρχία συνταγματικά σε ορισμένα κράτη-μέλη. Και αυτό έρχεται ακριβώς ως απάντηση σε ορισμένες προτάσεις που έρχονται από τις ξέλες που εκείνοι τις θεωρούν αιρετικές. Επομένως θα έλεγα ότι το θέμα είναι ευαίσθητο για όλα τα κράτη-μέλη. και έχοντας την εμπειρία των διαπραγματεύσεων στα, ε, στο Συμβούλιο Οικονομικών Υποθέσεων, γνωρίζω ότι ε, τα θέματα αυτά πρέπει να τίθενται και πρέπει να δίνει κανείς τις μάχες που χρειάζεται, αλλά ε, η δυνατότητα, επιμονή στην ε, κυριαρχία και στην ε, δυνατότητα κάθε κράτους μέλους να θέτει το φορολογικό του σύστημα ε, έχει οδηγήσει στο να χρειάζονται πάρα πολύ χρόνο οποιαδήποτε διαπραγμάτευση για βελτίωση των φορολογικών συστημάτων ή οποιοδήποτε συντονισμό. θα έλεγα ότι θα χρειαστεί ακόμα μία δεκαετία. Μην σας πω ότι οι περισσότεροι από εμά δεν θα είναι πια στα πράγματα όταν προοδεύσουμε στον τομέα αυτόν. Αυτή είναι η κατάσταση η οποία έχει σχέση και με τη δομή των θεσμικών οργάνων και τη λειτουργία τους. Η εναρμόνιση των φορολογικών συστημάτων ακούγεται όμορφα. Όμως, υπάρχουν διαφορετικά μοντέλα σε μεγάλα ε, και επιτυχημένα, αν θέλετε, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία έχουν καταφέρει με αυτόν τον τρόπο, με τη φορολογία που έχουν ε, δημιουργήσει, να μην έχουν ανεργία, να παρέχουν τις απαιτούμενες δημόσιες υπηρεσίες, έχουν δώσει απαντήσεις στις ανησυχίες των προβλημάτων των πολιτών τους. Επομένως, είναι λογικό να είναι απρόθυμα αυτά τα κράτη-μέλη να συζητήσουν μια ουσιαστική και μεγάλη μεταρρύθμιση των φορολογικών του συστημάτων. Τώρα θα μπορούσαμε να κάνουμε μια φιλοσοφική συζήτηση για το ποιες θα μπορούσαν να είναι οι αναλεκτικές ε, επιλογές αλλά ανταυτού θα σας έλεγα ότι με την υποστήριξη της ε, ε, Σλοβακικής Προεδρίας καταφέραμε να προοδεύσουμε και τελικά να υιοθετηθεί να υιοθετηθούν μέτρα όπως για παράδειγμα η οδηγία PIF για την καταπολέμηση διασυνοριακού ε, οικονομικού εγκλήματος η, επίσης η συμφωνία που, στην οποία καταλήξαμε ε, εχθές. Και αυτές οι πρόοδες σημειώθηκαν παρά το γεγονός ότι Ορισμένοι θεωρούσαν ότι τα θέματα αυτά επειδή άπτονται των φορολογικών συστημάτων δεν, για τα θέματα αυτά δεν θα μπορέσει να υπάρξει συμφωνία. Όσον αφορά τώρα την πρόταση της Γερμανίας, της Αυστρίας, της Τσεχίας για την αντίστροφη χρέωση, την ε, χρέωση του παραλήπτη των αγαθών, ε, ελπίζουμε ότι θα ελάβουμε τη σχετική πρόταση από την Κομισιόν ε, μέχρι τα Χριστούγεννα, πριν τα Χριστούγεννα. Η κυρία Τζέλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ. Επί Προεδρία σας επιτεύχθηκαν σημαντικά βήματα πρόοδου και θέλω να σας συγχαρώ. Είπατε κι εσείς ότι ψηφίσαμε ε, το πολιτισμό σημικό. Μάλλον ψηφίσαμε τα μηδέ κεφάλια της χρηματαγορίας, το MMF, ε, με μεγάλη πλειοψηφία σήμερα. Υπάρχουν σίγουρα αντικρώμενα συμφέροντα μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών. Θέλω να σας ευχαριστήσω εσάς και τη ομάδα σας, με και τον Κάμιλ Σάσκε. Νομίζω ότι ίσως να ήταν και μια από τις πιο δύσκολες διαπραγματεύσεις. Όλες είναι δύσκολες, αλλά αυτή πιο πολύ. Και νομίζω ότι ήταν καλό το ότι χθες έγινε το πρώτο νομοθετικό βήμα για την Ένωση Κεφαλαίου Αγορών. Αυτό που θέλω να πω εγώ τώρα είναι ότι η Προεδρία σας έχει αποτελέσματα και είναι θετικό αυτό. Η εμπειρία μου όμως μου λέει ότι πολλά από τα μικρότερα κράτη-μέλη δεν δείχνουν την, για το ίδιο θάρρος. Φαντάζομαι ότι συνομιλείτε με τους ε, συναδέλφους σας και ε, με τις επερχόμενες προεδρίες που πρέπει να σηκώσουν το γάντι ε, και ελπίζω να μην υπάρξουν προκλήσεις και εμπλοκές και να μείνουν εκτός κάποια θέματα, γιατί υπάρχουν σημαντικές οικονομικές και πολιτικές προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαι βέβαιη ότι έχετε επισημάνει αρκετές από αυτές. Χρειαζόμαστε όμω γρήγορη δράση. Θέλουμε ανάπτυξη οικονομική και θα πρέπει η Ευρώπη να πάψει να δείχνει τόσο κατακαιρματισμένη. Έχουμε την εντύπωση ότι το Συμβούλιο προσπαθεί όσο το δυνατό πιο γρήγορα ε, να αντιμετωπίσει, ε, αλλά δυσκολεύεται και πρέπει να προχωρήσουμε. Το τραπεζικό πακέτο θα είναι σίγουρα μια τέτοια πρόκληση και για τις επερχόμενες προεδρίες και είναι σημαντικό να ολοκληρωθεί το πακέτο να είναι πιο σταθερέ οι τράπεζε για να μπορούν να στηρίξουν για την ευρωπαϊκή οικονομία. Θέλω όμω να σα κάνω το εξή ερώτημα. Εσά σα ανησυχεί το επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η μείωση του δημόσιου χρέου σα ανησυχεί ε, στο BlackRock. Ε, η, έκθεση BlackRock δείχνει κάποια πράγματα που πρέπει να τα ανατρέψουμε σε τάσεις και τι θα πείτε στους Μαλτέζους και στους Εσθονούς για τις υπερχόμενες προεδρίες τους. Madam ja tiež eh, musím poďakovať za, za excelentnú spoluprácu a za hlavne schopnosť. Ευχαριστώ, κυρία Άτζιλ. Και με την ευκαιρία να σας ευχαριστήσω και για τη συνεργασία που είχαμε για την ε, οδηγία για τα ενημερωτικά δελτία. Και με χαρά διαπίστωσα επίσης ότι καταφέρατε να καταλήξετε σε συμφωνία με την ψηφοφορία σήμερα και στον τομέα της τίτλοποίηση. Καλό θα ήταν αυτό να είχε συμβεί λίγο νωρίτερα, γιατί τότε θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε τον τριμερή διάλογο, αλλά εντάξει. Ε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Οι συνάδελφοι από τη Μάλτα θα αναλάβουν τον φάκελο και σίγουρα θα προχωρήσουν τη διαπραγμάτευση. Τώρα επενδυτικά μία Καταφέραμε να συμφωνήσουν τα κράτη-μέλη, έτσι, όλα, έτσι ώστε να μην χρειαστεί να ε, χρησιμοποιήσουμε την αυξημένη πλειοψηφία, παρόλο που δεν ήταν όλοι 100% εικονοποιημένοι, Νομίζω όλοι αντιλαμβάνονται τη συμφωνία αυτής της συμφωνίας, τη σημασία αυτής της συμφωνίας. Νομίζω ότι όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αντιληφθεί ότι πρέπει να αποδείξουμε μετά το δημοψήφισμα για το Brexit ότι με ή χωρίς το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να, είμαστε, να επιτύχουμε την ολοκλήρωση της ε, Κεφαλαιακής Ένωσης. Γιατί το γεγονό ότι δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να ολοκληρώσουμε την Κεφαλαϊκή Ένωση ε, είναι μία από τι σημαντικότερε αδυναμίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση στον παγκόσμιο οικονομικό στίβο. Και αυτό δεν είναι ένα θέμα το οποίο μπορούμε να το κρύψουμε και να το ξεχάσουμε. Αναφερθήκατε επίση στο ζήτημα του δημοσίου χρέους. και των προσπαθειών που κάνουν τα διάφορα ε, κράτη για να χρηματοδοτήσουν τους εαυτού του. και προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματα της ποσοτική χαλάρωσης, το γεγονότος ότι τα επιτόκια είναι πάρα πολύ χαμηλά. Κάθε κράτο μέλος έχει την, στη διακριτική του ευχέρεια ε, να επιλέξει ποια μέτρα συγκεκριμένα θα ε, επιλέξει. ασκείται επίσης πίεση στα κρατικά ομόλογα στον τροπικό τομέα. Ε, αυτό είναι ένα θέμα που πιστεύω ότι δεν θα μπορέσουμε να λύσουμε πριν να λυθεί και να τελειώσει η ολοκλήρωση της Κεφαλαϊκής Ένωσης. Ε, σας μιλώ επίσης και ως υπουργό Οικονομικών μιας μικρής χώρας για να διασφαλίσουμε την πρόσβαση των χωρών όλων αυτών στις χρηματαγορές, της διεθνής θα πρέπει να φροντίσουμε ε, να τηρείται η δημοσιονομική πειθαρχία και το χρέος να είναι σε λογικά επίπεδα. Είναι ένα θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει πάρα πολλές φορές και η Κομισιόν συνεχίζει να ασχολείται με αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε ξανά στην ε, Επιτροπή ΕΚΟΝ σε σχέση και με αυτά που έλεγε η Σάρφος Γκίλ προηγουμένως και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ε, γιατί ολοκληρώσαμε ε, μαζί τον ε, φάκελο για τα αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να είστε και εσείς περήφανος για τη διαπραγματευτική σας ομάδα. Τώρα έχουμε ένα νέο πρόεδρο των ΗΠΑ, τον κύριο Τραμπ, ο οποίος όχι μόνο έχει, έχει εκλεγεί ο ίδιος, αλλά έχει και το Κογκρέσο μαζί του. Ε, ενδεχομένως, λοιπόν, θα προχωρήσει κάποια μέτρα όσον αφορά, ας πούμε, τον όσον αφορά τη φορολόγηση των ομίλων ε, στις Ηνωμένε ε, ε, Πολιτείες. Θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε γιατί αυτό μπορεί να έχει επίπτωση στην Ευρώπη. Ένα ενδεχομένως μπορεί να δημιουργήσει αύξηση του προϋπολογισμού και τη συμβολή του προϋπολογισμού καθώς επίσης και τροποποίηση των φορολογικών εισόδων σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, θα πρέπει τώρα στα πλαίσια του νέου προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να ληφθούν υπόψη όλα τα στοιχεία. Σκέφτεστε λίγο πώς μπορεί να προχωρήσουν τα πράγματα επίσης το θέμα του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, οποιαδήποτε και αν είναι η μορφή των σχέσεων που θα έχει το Ηνωμένο Βασίλειο με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχετε συζητήσει τις επιπτώσεις επίσης συζητήσαμε με το θέμα του φόρου ε, ε, των ε, χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και στο παρελθόν. Αλλά στο παρελθόν δεν καταφέραμε να επιτύχουμε οποιαδήποτε συμφωνία. Πιστεύετε ότι ε, ε, ότι υπάρχει περίπτωση ε, να προχωρήσετε στη συζήτηση έτσι ώστε να γίνει ένα παγκόσμιο πρότυπο και όχι μονάχα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απάντηση. Ορισμένα πράγματα έχουν απλουστευτεί και άλλα έχουν περιπλακεί περισσότερο είναι γεγονός ότι σε επίπεδο 10 χωρών ίσως δεν είναι πιο εύκολη η προσέγγιση, αλλά σίγουρα είναι καλύτερη όσον αφορά την ε, συνεργασία και την ε, ε, διευρυμένη συνεργασία όσον αφορά φορολογικά ζητήματα, το, τα θέματα ας πούμε των προτιμιστιακών καθεστώτων και ενδεχομένως την την, ε, από, την ε, ε, φυγή κάποιων εταιριών από χώρες οι οποίες δεν έχουν ευνοϊκό καθεστώς. Ναι, βεβαίως τα συζητούμε όλα τα θέματα αυτά, αλλά μας ενδιαφέρει κυριότερα ο πολιτικός χαρακτήρας του γενικότερου project. Συνάντησα τον κύριο Λεφέβρο ε, πριν από ένα μήνα περίπου στην ε, ε, Μπρατισλάβα και ήταν ο σύμβουλος του Προέδρου Ρίγκαν για θέματα φορολογικά πρέπει να σας πω ότι και αυτός περιμένει με μεγάλη ανυπομονησία το φορολογικό ε, καθεστώς ας πούμε στις Ηνωμένε Πολιτείες ε, το νέο ε, και ορισμένα από τα θέματα τα οποία ανέφερε και ορισμένα τα σχόλια, από τα σχόλια που έκανε για τις Ηνωμένε Πολιτείες ήταν ενδιαφέροντα, ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και στην συνάντηση που ανέφερα προηγουμένως στον ΟΣΑ συζητήθηκαν τα θέματα των φορολογικών πολιτικών ε, σε σχέση και με τις ε, νέες εξαγγελίες ε, της νέας κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με προστατευτισμό κτλ. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να περιμένουμε, να δούμε τη νέα κατάσταση. Ε, γιατί δεν τη γνωρίζουμε ακόμα. Θα πρέπει πάντως, ε, οπωσδήποτε, με επαγγελματισμό θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ε, οτιδήποτε προκύψει. Χωρίς να λησμονούμε ότι μας ενδιαφέρουν και οι εισαγωγές στις δικές μας αγορές. Όσον αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο, το σημαντικό είναι να παραμείνουμε ενωμένοι και να επιτύχουμε κοινέ θέσεις Ε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θέλουμε να πιέσουμε το Ηνωμένο Βασίλειο να επιταχύνει κάποιες ε, διαδικασίες. Θα πρέπει πολύ προσεκτικά να δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε δημοσιονομικά ζητήματα. Ε, ο Μάριο Μόντι είναι πάντα στην διάθεσή μας έτσι ώστε να βελτιώσει την ικανότητα αντίδρασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ε, πάντως εμείς ε, ε, ευχόμαστε τα καλύτερα, καλή επιτυχία στον κύριο Μπαρνιέ γιατί έχει μπροστά του δύσκολο έργο. Ευχαριστώ. Υπερβάνος Μπερές, τελευταία ομιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Στην πρώτη μου παρέμβαση θα έπρεπε να σας είχα συγχαρώ βεβαίως ε, γιατί κάνατε αυτό το άτυπο συμβούλιο στα πλαίσια του οποίου ε, συζητήσατε με τους συναδέλφους σας ε, στο θέμα της ελάχιστης αποζημίωσης ανεργίας και επίσης την συζήτηση για την δημοσιονομική ικανότητα ε, και τα aggregated standards. Ε, φαντάζομαι ότι τα θέματα αυτά θα τα περάσετε και στην ε, Προεδρία της Μάλτας. Και το θέμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε σχέση και με αυτό που έλεγε ο κ. Μπερναρλάνγκη Λάγκε προηγουμένως. Ε, ξέρω ότι στο Συμβούλιο ΔΕΗ τα συζητάτε τα θέματα αυτά, αλλά χρειαζόμαστε, ξέρετε, ε, την υλοποίηση αυτής της ε, Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και είμαστε λίγο απογοητευμένοι από τα αποτελέσματα. δεν θεωρείτε ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε προς ενισχυμένη συνεργασία και κατά αυτή την έννοια πρωτοβουλίες που είχαν ε, αναλυφθεί από τις ε, προεδρίες της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας θα πρέπει να προωθηθούν ε, περισσότερο έτσι ώστε να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε μια ευρωπαϊκή εισαγγελία του έστω και σε εμβριακή κατάσταση η οποία θα μπορέσει να αντιμετωπίσει θέματα μεγάλης εγκληματικότητας και οπωσδήποτε και τρομοκρατίας. Um, uh, Κυρία Θα ήθελα να σας πω ότι εμείς από την αρχή προσπαθήσαμε να δούμε το θέμα της ολοκλήρωσης της νομισματικής ένωσης με ραλιστικό τρόπο. Δεν θέλαμε να φανούμε αφελείς. Πάντοτε μπορεί κανείς να ονειρεύεται και να ελπίζει για το τι θα προκύψει ε, μετά από 10 χρόνια, πώς θα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από 10 χρόνια. Είπατε για κάποιες πρωτοβουλίες. Εμείς επιλέξαμε την ε, επιστολή ως μέσο, επιστολή της Προεδρίας. Θα αναφέρουμε όλες τις πρωτοβουλίες και θα σας πούμε επίσης ποια ήταν η ατμόσφαιρα και η φύση των συζητήσεων και των μεταξύ των και πολιτικών πρωτοβουλειών που πήραμε. Θα διαβιβαστεί στον ε, πρόεδρο Σούλτς αυτή η επιστολή, φυσικά. Και ελπίζω ότι με τον τρόπο αυτό ίσως ε, θα δώσουμε και κάποια έμπνευση για τους συντάκτες της ε, Λευκής Βίβλου που θα πρέπει να δημοσιοποιήσει η Κομισιόν του χρόνου το Μάρτιο. Ίσως και συμπεριληφθεί και στον οδικό χάρτη της Μπρατισλάβα που συμφώνησαν να εφαρμόσουν οι ηγέτες μας το καλοκαίρι. Και η Μάλτα θα πρέπει να ανταποκριθεί, ε, να αντιδράσει σε αυτό το οδικό χάρτη που θα, συγγνώμη, σε αυτό τη λευκή βιβλίο που θα δημοσιοποιήσει η Κομισιόν το Μάρτιο. Ελπίζω όμως να είναι πηγή και να μην φοβήσει κανέναν. Γιατί οι πραγματικότητες που θα περιγράφει μπορεί να μην είναι πάντοτε ευχάριστες για όλους. Εσείς μιλήσατε για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το Γραφείο Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Συμφωνώ, ναι, δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Απλά θέλω να σας υπενθυμίσω πως με δική μας πρωτοβουλία, Επιτρόπος Γιούροβα, δύο φορές μίλησα στο ΕΚΟΦΗΝ, κάτι ασυνήθιστο, και είδαμε τα θέματα φοροαποφυγής, φοροαπα... Ε, φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής ε, και απάτης ε, με το ΦΠΑ. Χάνονται εκατομμύρια, δισεκατομμύρια. Γιατί υπάρχει μεγάλη συνεργασία, διαπλοκή μεταξύ των τρομοκρατικών και εγκληματικών κυκλωμάτων. Εμείς ε, καταλήξαμε σε συμπεράσματα και μάλιστα μέχρι που καταφέραμε να πείσουμε και ορισμένα κράτη-μέλη που δεν είχαν θετική άποψη για το γραφείο του Ευρωπαϊκού Αγγελίου. Αν δεν απατώμε το Τζάι θα τα συζητήσει αύριο αυτά τα θέματα το Συμβούλιο Εσωτερικών και Δικαιοσύνη. Αυτά είχα να πω για το θέμα. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ Πέτερ, ήταν πολύ καλή αυτή η ανταλλαγή απόψεων και για μια ακόμη φορά σας συγχαίρω για την πολύ επιτυχημένη Προεδρία, τα πολύ μεγάλα επιτεύγματα όλα όσα αναφέρατε και σε ό,τι αφορά ε, τους για τα ΜΒ κεφάλαια να δώσετε συγχαρητήρια και για τη δημοσιονομική ικανότητα ηγηθήκατε αυτών των συζητήσεων και ελπίζω ότι και με τη συμβολή του Κοινοβουλίου να παραμείνει στην ατζέντα αυτό το θέμα γιατί είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον της ΟΝΕ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Επόμενη συνεδρίαση την προσεχή Δευτέρα, αγαπητοί συνάδελφοι. Κύριος Κάζιμιρ, καλά Χριστούγεννα, ευχαριστώ για τη συνεργασία.